Οι πολιτικές είναι αυτό το οποίο θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και για να το καταφέρουν θα πρέπει να διέπονται από φιλοδοξία αλλά και από ρεαλισμό. Δεδομένου λοιπόν του κεντρικού ρόλου που παίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκέ πολιτικέ είναι κατάλληλε για του Ευρωπαίου πολίτε, δεν θα μπορούσα να βρεθώ σε καλύτερο χώρο προκειμένου να συζητήσω μαζί σα τα θέματα τα οποία επιλέξατε. Όπω είπατε, τα δύο θέματα αυτά είναι κεντρικά τη σήμερον ημέρα. Πρώτα θα μιλήσω λοιπόν για την εξέλιξη της οικονομικής προοπτικής και της αβεβαιότητας και στη συνέχεια θα μιλήσω για το ρόλο της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το ρόλο που μπορεί να παίξει και η δημοσιονομική πολιτική. Μίλησα ήδη για την αβεβαιότητα. Πράγματι αυτό χαρακτηρίζει την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Κάτι το οποίο βέβαια κάνει ακόμα πιο δύσκολο το δικό μας τον ρόλο και το δικό σας φυσικά. Οπότε ας κοιτάξουμε λιγάκι τις οικονομικές προοπτικές. Όπως είπα, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Λοιπόν, τα τελευταία νέα που έχουμε όσον αφορά τα εμβόλια, προφανώς και δείχνουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Οι τελευταίες έρευνες που έχουν γίνουν για την περίπτωση του κορονοϊού και τα εντατικά μέτρα περιορισμού ήδη ε, ελήφθησαν για να αντιμετωπιστεί η αβεβαιότητα και αποτελούν μεγάλη πρόκληση για την Ευρωζώνη στο σύνολό της. Υπάρχει μία ανάκαμψη η οποία όμως δεν είναι ίδια παντού και οι διάφορες έρευνες δείχνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη ε, πέρασε σε δυναμία κάπως το τελευταίο τρίμηνο. Και φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο βαραίνει ιδιαίτερα κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών. για λόγους που φυσικά όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά είναι ιδιαίτερα ευάλωτος ο τομέας αυτός εξαιτίας των ε, φυσικών αποστάσεων που πρέπει όλοι να τηρούμε μεταξύ μας. Ο δείκτης, ο PMI, όσον αφορά την Ευρωζώνη, δείχνει ότι ενώ η μεταποίηση βελτιώνεται, οι δραστηριότητες στις υπηρεσίες ε, επιβραδύνονται αισθητά τον Οκτώβριο. Και βέβαια με άνηση κατάσταση, κάτι το οποίο το βλέπουμε σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, ε, κυρίως για εκείνες που εξαρτώνται κατά πολύ από τα ταξίδια και τον ε, τουρισμό. Μέχρι τώρα τα μέτρα των κυβερνήσεων στήριξης έχουν προστατεύσει τα νοικοκυριά από την ανεργία και από την απώλεια εισοδήματος. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι η ανεργία δεν αυξήθηκε πολύ σε κάποιες χώρες. Οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί μέσα σε αυτό το πλαίσιο βεβαιότητας στο οποίο ζούμε, γιατί η πανδημία απειλεί τις θέσεις απασχόλησης και τις οικονομικές προοπτικές του κόσμου. Είναι χαμηλή η ζήτηση, υποτονική και η κερδοφορία, κάτι το οποίο επηρεάζει και τις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις θα εξακολουθήσουν να διστάζουν να δεσμεύσουν χρήματα σε επενδύσεις μακροπρόθεσμα, όσο εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα για το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία και πώς, όπως επίσης και για το πώς θα προχωρήσουν τα εμβόλια και πώς επιτυχή θα είναι. Συνολικά λοιπόν η οικονομία στην Ευρωζώνη αναμένεται να επηρεαστεί σοβαρά από την ε, μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων και την αντατικοποίηση των περιορισμών. Κάτι το οποίο οδηγεί σε καθοδικούς ε, κινδύνους όσον αφορά την οικονομική προοπτική. Η αδυναμία λοιπόν στην οικονομική δραστηριότητα από τότε που ξεκίνησε η πανδημία αντικατοπτρίζεται επίσης και στις εξελίξεις όσον αφορά τον πληθωρισμό. Οι χαμηλές τιμές ενέργειας και η προσωρινή μείωση του φόρου προσθέμενης αξίας στην Γερμανία επηρεάζουν τον πληθωρισμό. Όμως η αδύναμη ζήτηση κυρίως στον τουρισμό και στους τομείς που έχουν να κάνουν με ταξίδια όπως ε, επίσης και η κατάσταση στις παραγωγικές αγορές οδηγούν σε μεγαλύτερη πίεση προς τα κάτω. Αναμένουμε συνεπώς ότι ο μετρούμενος πληθωρισμός θα παραμείνει αρνητικός μέχρι τις αρχές του 2021. Ο ρόλος κλειδί της νομισματικής πολιτικής συνεπώς είναι να προστατεύσει και να προσφέρει ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης σε όλους ε, τους τομείς και σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης και να στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα και να διασφαλίσει την ε, σταθερότητα τιμών μεσοπρόθεσμα. Όταν λοιπόν ε, σκεφτόμαστε ευνοϊκέ συνθήκε χρηματοδότηση, αυτό που έχει κυρίω σημασία δεν είναι τόσο το επίπεδο τη χρηματοδότηση, αλλά η διάρκεια των ε, πολιτικών στήριξή τη. Έτσι λοιπόν η διατήρηση ευνοϊκών συνθήκων χρηματοδότησης χρειάζεται για να στηριχθεί ο κόσμος να μπορεί να δαπανά, να υπάρχει ροή χρήματος και να αντισταθμίσονται οι απολύσεις. Έτσι λοιπόν το Δικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει τις εισερχόμενες πληροφορίες, κυρίως όσον αφορά το νέο στάδιο προβολών του Δεκεμβρίου των Επιρρογνωμόνων και έτσι θα μπορέσουμε να επαναξιολογήσουμε τις οικονομικές προοπτικές και να αξιολογήσουμε και το ισοζύγιο κινδύνων. Βάσει λοιπόν αυτή τη επικαιροποιημένη αξιολόγηση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναπροσαρμόσει καταλήλω τα μέσα που διαθέτει, προκειμένου να αποκριθεί στην κατάσταση όπως αυτή εξελίξεται και να διασφαλίσει ότι οι συνθήκε χρηματοδότησης παραμένουν ευνοϊκές, ώστε να στηρίξουν την οικονομική ανάκαμψη και να αντισταθμίσουν την αρνητική επίδραση της πανδημίας στην πορεία του πληθωρισμού και στη σύγκληση του πληθωρισμού σύμφωνα με την δέσμευσή του για συμμετρία. Τώρα, γνωρίζετε ε, τα διάφορα προγράμματά μας. Το ΠΕΠ πρώτα απ' όλα, το οποίο είναι πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού πανδημίας, που έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό στο σημερινό πλαίσιο και μπορεί να προσαρμοστεί για να αντιδράσει στις εξελίξεις όσον αφορά την πανδημία. Συνεπώς, τα προγράμματά μας αγορά στοιχείων ενεργητικού θα είναι και τα κύρια μέσα που διαθέτουμε για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Αντιδράσαμε γρήγορα και δυναμικά στο πρώτο κύμα της πανδημίας για να βοηθήσουμε τις οικονομίες της Ευρωζώνης με προγράμματα σχεδιασμένα για να αντιμετωπιστεί ο τριγμός της πανδημίας με τα κατάλληλα μέσα. Τα μέτρα μας ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικά γιατί σταθεροποίησαν τις αγορές και ενίσχυσαν την οικονομική δραστηριότητα. Βοήθησαν δηλαδή να αντισταθμιστεί η καθοδική πορεία της οικονομίας λόγω της πανδημίας. Θα αντιμετωπίσουμε λοιπόν και το τωρινό στάδιο της πανδημίας με την ίδια προσέγγιση και την ίδια αποφασιστικότητα. Επιτρέψτε μου τώρα να στραφώ στο δεύτερο θέμα που επιλέξατε και που είναι η σύνδεση ανάμεσα στη δημοσιονομική και την νομισματική πολιτική. Η απάντηση στην κρίση προς το παρόν έχει δείξει πώς αμοιβαία. Η νομισματική και η δημοσιονομική πολιτική μπορούν να ενισχύσουν η μία την άλλη. Για την νομισματική πολιτική, σας εξήγησα προηγουμένως, είναι ζωτική σημασία να διασφαλίσουμε ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης για ολόκληρη την οικονομία. Συγχρόνως, η δημοσιονομική πολιτική έχει να παίξει σημαντικό ρόλο, ενισχύοντας την ζήτηση, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και ενισχύοντα ε, επίσης τις δυνατότητες που έχουν οι οικονομίες μας. Η δημοσιονομική πολιτική, από την άλλη μεριά, έχει σημαντικό ρόλο για τρεις λόγους κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, κινητοποιεί την οικονομία γρήγορα, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Δεύτερον, η δημοσιονομική πολιτική έχει και τομεική διάσταση, κάτι το οποίο δεν έχει η νομισματική πολιτική. Και τρίτον, κάποια από τα εργαλεία πολιτικής, για παράδειγμα εγγύσεις πιστώσεων, είναι κάτι καθαρά δημοσιονομικό από τη φύση του. Σήμερα οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης έχουν υιοθετήσει δημοσιονομικά μέτρα για πάνω από 4% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης για το 2020 και στηρίζουν με ρευστότητα την οικονομία και με αυτοματοποιημένους σταθεροποιητέ. Οι δημοσιονομικές απαντήσεις λοιπόν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικές διότι συγκρατήθηκε η ανεργία, υπήρξαν εγγύσεις δανείων, ε, απασχόληση και χάθηκαν λιγότερες επιχειρήσεις. Και τα μέτρα αυτά τα δημοσιονομικά συμπληρώθηκαν και αποστήριξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα λεγόμενα δίκτυα ασφάλειας που ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη αυξήθηκε η ζήτηση, διευκολύνθηκε η πρόσβαση σε πιστώσεις για επιχειρήσεις κυρίως. Αυτά είναι μέτρα τα οποία ενισχύουν και την αποτελεσματικότητα της νομισματικής μας πολιτικής. Ενώ λοιπόν τα δημοσιονομικά μέτρα τα οποία λήφθησαν για απάντηση στην πανδημία πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά από τη φύση τους, η ασθενή ζήτηση και οι κίνδυνοι μιας καθυστερημένης ανάκαμψης χρειάζονται συνεχή στήριξη από τις εθνικές ε, δημοσιονομικές πολιτικές και χρειάζεται συντονισμός και πρέπει με κάθε τρόπο να αποφύγουμε τα φαινόμενα κατακριμνισμού. Οι δημόσιες επενδύσεις μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική ανάπτυξη στη σημερινή κατάσταση. Μέσα σε ένα περιβάλλον διευκολυντικής ε, νομισματικής πολιτικής, οι δημόσιες επενδύσεις έχουν γρήγορα αποτελέσματα και συμπεριλαμβάνουν ε, και τις επιπτώσεις που έχουν ε, στις γειτονικέ χώρες. Όταν υπάρχει μεγάλη βεβαιότητα, οι δημόσιες επενδύσεις ενισχύουν την εμπιστοσύνη και λειτουργούν και σαν ε, πολλαπλασιαστής. Αυξάνοντας την εμπιστοσύνη, οι δημόσιες επενδύσεις επίσης δημιουργούν και καλύτερο πλαίσιο για επενδύσεις από τους ιδιωτικούς φορείς. Συγχρόνως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα και οι επιπτώσεις στα δημοσιονομικά των χωρών εξαρτώνται από την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων και από την παραγωγικότητα του δημοσίου κεφαλαίου. Οι δημόσιες επενδύσεις λοιπόν και οι μεταρρυθμίσεις κυρίως μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για να αντιμετωπιστούν τέτοιες δυσκολίες όπως είναι η η ψηφιοποίηση, χρειάζονται μια συνολική ανάκαμψη χωρίς να ξεχαστεί κανείς. Κανένας δεν πρέπει να μείνει σε απομόνωση. Πρέπει να συνδυάσουμε τις μεταρρυθμίσεις με ε, τα κίνητρα για επενδύσεις, γιατί έτσι θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η ανάκαμψη. Και τα δύο μαζί θα διαμορφώσουν το μέλλον των οικονομιών μας και θα διασφαλίσουν ότι οι οικονομίες μας προσαρμόζονται στη νέα κανονικότητα, η οποία θα υλοποιηθεί όταν ξεπεράσουμε την ε, αναζωγόνηση αυτή της πανδημίας. Για αυτούς τους λόγους, το πακέτο Next Generation EU πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί χωρίς καθυστέρηση. Είναι ζωτική σημασία σε αυτό. Τα επιπλέον ε, πακέτα ε, πόρων θα διευκολύνουν επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές, κυρίως στις χώρες εκείνες της Ευρωζώνης που δεν έχουν πολλά δημοσιονομικά περιθώρια. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε και διακανονισμούς για να επιτρέψουμε αποτελεσματικές δαπάνες των κονδυλίων αυτών. Γι' αυτό και χαίρομαι για την πρόσφατη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία όσον αφορά την χρήση τη δημοσιονομική αυτή στήριξη από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σήμερα περισσότερο σημαντικό από ποτέ, τόσο για την νομισματική όσο και για τη δημοσιονομική πολιτική, να συνεχίσουν να συνεργάζονται χέρι-χέρι, όπω έχει γίνει μέχρι σήμερα. Οι συνθήκε διασφαλίσουν ότι αυτό μπορεί να γίνει σεβόμενη πλήρω την εντολή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την ανεξαρτησία τη. Και καταλήγω λέγοντα ότι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρίση μέχρι σήμερα ήταν εντυπωσιακή, αλλά και ιδιαίτερα αποτελεσματική συγχρόνως. Μπήκαμε στο δεύτερο στάδιο της κρίσης και πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα και δέσμευση να δίνουμε αποτελέσματα, να φέρουμε αποτελέσματα για ε, τους λαούς της Ευρώπης. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, περίπου όλοι σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, που σίγουρα γνωρίζετε, ζητούν τέτοια δράση από τη δικιά μας την πλευρά. Όπως είπα και στην εισαγωγή μου, να διασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές που διαμορφώνουμε σήμερα μας επιτρέπουν να τα καταφέρουμε. Όπως και ο Γιώχαν Βόλφκαν Φανγκέτε είπε, στα αγγλικά τουλάχιστον, δεν το είπε στα αγγλικά εκείνο, εγώ το λέω στα αγγλικά, λέει η κυρία Λαγκάρτ, σε το βασίλειο των ιδεών όλα εξαρτώνται από τον ενθουσιασμό. Στον πραγματικό κόσμο όλα βασίζονται στην επιμονή. Πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you very much for this insight. Ευχαριστώ πολύ για αυτά που μας είπατε. Θα ξεκινήσουμε τώρα την περίοδο ερωτήσεων-απαντήσεων. Θα δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές θα έχουν δύο λεπτά ο καθένας. Παρακαλώ να το χρόνο σας και μετά πρόεδρε Λεγκάρντ θα μπορείτε να απαντήσετε και θα έχετε τρία λεπτά για την απάντησή σας, χωρίς να περιμένετε για μένα να σας δώσω το λόγο, ώστε να εξοικονομήσουμε χρόνο και να αποφύγουμε προβλήματα συνδέσεων. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Μάρκους Φέρμπερ από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και χαίρομαι που έχετε βολευτεί ήδη τόσο καλά στην Φραγκφούρτη και που απαγγέλλετε και γκέτε. Δύο ερωτήσει έχω να κάνω. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην εποχή του κορονοϊού θα πρέπει να παραμείνει ενεργή. Το Δεκέμβριο Ε, ρυθμίζεται και υπολογίζουμε ότι υπάρξει αύξηση του ΠΕΠΣ. Και εδώ τίθεται θέμα νομιμότητας του ΠΕΠΣ. Και το δικαστήριο έχει επιβεβαίωση ότι είναι νομικά βάσιμη η δράση ως τώρα του ΕΚΤ σε ό,τι αφορά τα μη ε, επιλεκτικά μέτρα, σε ό,τι αφορά τα ανατολικά όρια στις επενδύσεις από πλευρά της ΕΚΤ και σε ό,τι αφορά τις κλίδες κεφαλαίου. Με το ΠΕΠ, λοιπόν, η ΕΚΤ έχει τη μέγιστη ε, ευελιξία σε ό,τι αφορά α, τα, τα όρια. Συνάδει, λοιπόν, το α, ΠΕΠ με την απόφαση του δικαστηρίου. Και δεύτερη ερώτηση. Το σύστημα πληρωμών ΚΑΓΚΙ 2. και σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που υπήρχαν με τους υπολογιστέ, οι επιπτώσεις που υπήρχαν ε, στις πληρωμές, οι οποίες, ε, τα οποία επιλύθηκαν, προβλήματα που επιλύθηκαν στο Σαββατοκύριακο. Έχετε, είστε αρμόδιοι ε, και για τα θέματα εποπτείας τραπεζών και σε αυτό συγκαταλέγεται και το θέμα της λειτουργία ε, λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων. Ποια είναι λοιπόν τα συμπεράσματα τα οποία μπορείτε να εξαγάγετε από τα υπολογιστικά αυτά προβλήματα που προέκυψαν από το KKG2. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ η απάντηση της κυρίας Λαγκάρτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις δύο αυτέ. αυτές και ναι, πάντα πρέπει να πω ότι χαίρομαι που βρίσκομαι στη Φραγκφούρτη σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος. Να παρατηρήσω το εξή. Η απόφαση στην οποία αναφέρεστε εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογή ρητά οποιαδήποτε προγράμματα έκτακτα τα οποία ήταν υπό εξέλιξη την εποχή που ήταν υπό αναθεώρηση το πρόγραμμα και το θυμάμαι αυτό, το διάβασα ξεκάθαρα στην απόφαση. Να πω το εξής. Το πρόγραμμα αγορών ε, κατεπίγουσας ανάγκης για την πανδημία όντως καταστρώθηκε υπό εξαιρετικές συνθήκες για να αντιμετωπιστεί η πανδημία και οι επιπτώσει της στην οικονομία μας. Άρα, ω εκ τούτου είναι πάρα πολύ στοχευμένο. Στοχευμένο κατ' και προσωρινής φύσεως. Έχετε τι λοιπόν δράση. Καταρχάς, να εξασφαλίσει ότι θα υπάρξει σταθερότητα στις αγορές προκειμένου να δοθεί χρηματοδότηση και κατά δεύτερον έχει και μία νομισματική λειτουργία. Δεδομένων λοιπόν των ε, έκτακτων συνθήκων που επικρατούσαν τότε ήταν κάτι απαραίτητο. Ήταν απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ένας τριπλός μηχανισμός ευελιξίας σε ό,τι αφορά τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αγοραζόντουσαν, τα οποία ήταν διαφορετικά από τα παραδοσιακά προγράμματα του παρελθόντος, ευελιξία σε ό,τι αφορά το χρόνο, άρα έπρεπε να γίνει front-loading των αγορών που γίνοντουσαν και ευελιξία σε ό,τι αφορά ε, τις δικαιοδοσίες, γιατί προφανώς για να επανέλθει η σταθερότητα η δημοσιονομική που επιθυμούσαμε στις αγορές έπρεπε να συντρέχουν αυτές οι τρεις ε, πτυχές, αυτές οι τρεις πτυχές της ευελιξίας που χρησιμοποιήθηκαν από την αρχή του προγράμματος. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι κοιτώντα ε, ότι αυτές οι αγορές σαν σε τεμηνιαίο επίπεδο, η ευελιξία η οποία ήταν απαραίτητη στην αρχή ήταν λιγότερο απαραίτητη στην πορεία, γιατί σημειώσαμε ε, μεγάλη επιτυχία. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον πρώτο στόχο, σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, και από ό,τι φάνηκε, από την απόδοση στον ευρωπαϊκό χώρο και σε ό,τι αφορά και τα αποτελέσματα στον επιχειρηματικό κόσμο. Δεδομένη λοιπόν της έκτακτης ε, φύσης και του προγράμματος και των συνθήκων, αυτές οι πτυχές ευελιξίας, οι οποίες ήταν πάρα πολύ απαραίτητες στην αρχή και λιγότερο τώρα, ήταν ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του προγράμματος και ήταν ε, απαραίτητες και πρέπει να πω ότι επιτέλεσαν το σκοπό τους σε ό,τι αφορά την επιτεύξη της σταθερότητας στον ε, ε, χώρο του ευρώ, της ευρωζώνης. Κατά δεύτερον, η δεύτερη ερώτηση για το σύστημα πληρωμών και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Με ανησυχούν. Γιατί, όπως είπατε κι εσείς, η αποτελεσματική και ταχεία διεξαγωγή πληρωμών μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων αποτελεί μια πολύ σαφή λειτουργία για την οποία είναι αρμόδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε μια αναθεώρηση και του προβλήματο αυτό που παρουσιάστηκε, αλλά και προηγούμενων προβλημάτων. Έχουν παρουσιαστεί τέσσερα άλλωστε του τελευταίους μήνε. Σε ό,τι αφορά το System Target 2. Θα γίνει λοιπόν αυτή η έρευνα, η σχετική, χωρίς ε, καμία μα, καθυστέρηση και χωρίς καμία επίοικια, γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς ποια είναι η αιτία, τι πρέπει να διορθώσουμε, γιατί υπήρξε αυτή η διακοπή, ήταν ανθρώπινο σφάλμα, ήταν ε, διακοπή ηλεκτρικού. Δεν πιστεύω ότι ήταν ανθρώπινο σφάλμα, αλλά, ε, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να εξετάσουμε με ανοιχτό πνεύμα το τι συνέβη για να βρούμε την πραγματική αιτία και να την τερθώσουμε. Και προφανώς ε, το Eurosystem γενικότερο, γιατί αυτά τα ζητήματα παρουσιάζονται γενικά στο Eurosystem, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και προφανώς υπάρχει μεγάλη διασύνδεση σε ό,τι αφορά το σύστημα πληρωμών, αλλά όλο το σύστημα Eurosystem ε, θα βεληθεί από τα συμπεράσματα που θα εξάγαμε από τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν με πλήρη διαφάνεια για να έχουμε πραγματικά δομές και υποδομές που θα είναι διαφανείς και θα λειτουργούν εύρυθμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα να δώσω το λόγο στον ε, Χουάν Φερνάνδες από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. We can hear you. Okay, thank you, thank you. Σας ακούμε, ναι, μάλιστα, ευχαριστώ. Γιώνας Φερνάνδες. Καλώ ορίσατε, κυρία Λαγκάρτ. Θα μιλήσω ισπανικά. Τις τελευταίες εβδομάδες ακούσαμε για την σχέση ανάμεσα στην νομισματική και τη δημοσιονομική πολιτική. Αναφερθήκατε και εσείς στο δεύτερο τμήμα της παρέμβασής σας. Τις τελευταίες εβδομάδες φάνηκε ε, με την ανακοίνωση για τα εμβόλια να μειώνεται η αβεβαιότητα και η περίοδος κατά την οποία θα πρέπει να συνεχίζονται οι περιορισμοί. Τις τελευταίες ημέρες όμως ακούσαμε την θέση των κυβερνήσεων της Σλοβενίας, της Ουγγαρίας, ε, Πολωνίας κτλ. που αναφέρθηκαν στην δυνατότητα να περιμένουμε τον προπολογισμό Next Generation EU. Εσείς Πιστεύετε ότι έτσι θα αυξηθεί η αβεβαιότητα, οπότε θα κληθείτε κι εσείς ανάλογα να πάρετε αποφάσεις στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο για αυτήν την συνεδρίαση. Οι προβλέψεις είναι, όσον αφορά τον πληθωρισμό είναι πολύ μακριά από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. στο ίμιση τουλάχιστον της εντολής σας δεν θα έχει επιτευχθεί ο στόχος της ΕΚΤ. Οπότε τις επόμενες εβδομάδες μπροστά θα έπρεπε να πάρετε πιο φιλόδοξα μέτρα ώστε να στηρίξετε ε, αυτή την περίοδο ε, αβεβαιότητας και να προσπαθήσετε να πλησιάσετε το στόχο σας. Ευχαριστώ. Πολύ θα ήθελα να μπορούσα να σας απαντήσω αλλά δεν άκουσα καθόλου την αγγλική διερμηνία, λέει η κυρία Λαγκάρτ. Θα τα πω στα αγγλικά, λέει ο κύριος Φερνάντες. Εντάξει, θα τα πω και στα αγγλικά. Με ακούτε? Σας ακούμε κύριε Φερνάντες. Ωραία, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, έλεγα η πρώτη μου ερώτηση ήταν ότι όπως ξέρετε ε, κάποιες χώρες αποφάσισαν στο Συμβούλιο να μπλοκάρουν τον προπολογισμό για το New Generation EU. Στη, στο δεύτερο τμήμα της ομιλίας σας, εσείς αναφερθήκατε στη σχέση ανάμεσα στη νομισματική και την δημοσιονομική πολιτική. Και ήθελα να σας ρωτήσω για αυτή τη νέα βεβαιότητα που προκύπτει όσον αφορά ε, το χρόνο που θα υλοποιηθεί ο νέος αυτός προϋπολογισμός. Και η άλλη μου ερώτηση είχε να κάνει με την νομισματική πολιτική, γιατί ο πληθωρισμός κάθε άλλο παρά κοντά στο στόχο βρίσκεται και με τις σημερινές προβλέψεις τουλάχιστον για το ίμιση της θητείας σας δεν θα συμμορφωθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τον κύριο στόχο της, την κυρία εντολή τη. Οπότε μήπως επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να ληφθούν νέες αποφάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο. για να περιοριστεί μέρος της αβεβαιότητας τουλάχιστον που προκλήθηκε εξαιτία των τελευταίων συμβάντων στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη που σας ανάγκασα να επανελάβετε την ερώτησή σας. Ίσως θα έπρεπε θα βάλω το γαλλικό κανάλι, δεν ξέρω. Τέλο πάντων, τώρα ναι, κατάλαβα την ερώτησή σα. Λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο τμήμα, που δεν είναι πραγματικά ερώτηση, αλλά τέλο πάντων μου δίνει την ευκαιρία να επαναλάβω ότι το Next Generation EU και οι προσπάθειες που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν πολύ σημαντικά στοιχεία της απάντησης στην κρίση. Σε πανευρωπαϊκή βάση βέβαια πολύ σημαντικό στοιχείο των δημοσιονομικών ε, και νομισματικών μέτρων της σύνδεσης αυτής της δημοσιονομικής με την νομισματική διάσταση. Κάτι πάρα πολύ θετικό. Οπότε όσο πιο γρήγορα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, το Next Generation EU και το RFF, προκειμένου να καθυσυχαστούν οι ανησυχίες τόσο το καλύτερο. Ελπίζω λοιπόν το Σεβούλιο να τα καταφέρει. Και να γίνει αυτό σύντομα. Τώρα για τη δεύτερη ερώτησή σας. Όταν κοιτώ τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το οποίο περιέγραψα απαντώντας στην προηγούμενη ερώτηση που είναι από την νομισματική άποψη και λαμβάνοντας υπόψη την εντολή σταθερότητας τιμών, νομίζω ότι τα κατάφερε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα κατάφερε χρησιμοποιώντας δύο ε, στοιχεία κλειδί. Το ένα είναι το πρόγραμμα αγοράς ενεργητικού ΠΕΠ, το έκτακτο, και το άλλο είναι το TLTRO, που είχε σαν στόχο να ενθαρρύνει τις τράπεζες να συνεχίσουν να δανείζουν στην οικονομία. ακριβώς για να μπορούμε να επωφεληθούμε και από χαμηλά επιτόκια. Έτσι νομίζω αποκαταστήθηκε εν μέρη η σταθερότητα και δημιουργήθηκαν ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης για τη στήριξη της ανάκαμψης της οικονομίας, το είδαμε αυτό το Μάιο και τον Ιούνιο εξάλλου, και επίσης ε, πετύχαμε και τη δέσμευσή μας για τη σταθερότητα τιμών. Αν δείτε τώρα τι λένε οι προβλέψεις των επιρογνωμόνων για το τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, από τις αποφάσεις μας του Μαρτίου δηλαδή μέχρι τα τέλη του 2022, δεν πρόκειται μόνο για το 1,3% παραπάνω που βάζουμε στο τραπέζι ή τι κάνουμε για τον πληθωρισμό. Όλα αυτά τα μέσα μέτρησης δείχνουν ότι εμείς κάναμε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουμε. Βέβαια, πρέπει να δούμε και τι θα είχε συμβεί αν δεν είχαμε δράσει. Αυτό βέβαια δύσκολα μπορεί κανείς να το αποδείξει, αλλά από τις μελέτες τουλάχιστον ε, τις οποίες διεξάγουν οι ε, συναδελφοί μου, αυτό ακριβώς φαίνεται. Ότι τα καταφέραμε με το πρώτο κύμα, φέραμε αποτελέσματα, τώρα είμαστε στο δεύτερο κύμα και θα συνεχίσουμε. Ακριβώς το ίδιο. Και τον Οκτώβριο, στη συνεδρίαση του Δικητικού Συμβουλίου, το είπα ότι θα υπάρξει επαναστάθμιση των ε, μέτρων που παίρνουμε εφόσον χρειάζεται. Να δώσουμε το λόγο στο Λίσ Γκαρικάν από το ΡΙΝΙΟΥ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και χαίρομαι που είσαστε εδώ, κυρία Λαγκάρτα. Πριν από κάποιες ημέρες στο Ευρωπαϊκό Ιούλιο. είχαμε ένα πάνελ εμπειρογνωμόνων για να κάνουμε μια συζήτηση για φέτος. Και ο κ. Σασάτ, τον οποίο γνωρίζετε καλά, μίλησε για τους ε, υπερβολικούς κινδύνους που έχουμε στο PCB ό,τι αφορά το πρόγραμμα αγορών ενεργητικού της πανδημίας, ε, το οποίο συστάθηκε, σας συγχαίρω γι' αυτό και λειτουργήσε πολύ καλά σε ό,τι αφορά τη σταθεροποίηση των ε, ε, οικονομικών αγορών, αλλά το θέμα λοιπόν αυτό έχει να κάνει και με τις διάφορες χώρες, με δημοσιονομικά, όχι νομισματικά μέσα. Αν λοιπόν μία χώρα δεν συμπεριφέρεται όπως πρέπει, μπορούμε να την διορθώσουμε με πολλούς τρόπους. Και κάποιες χώρες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, αρνούνται να χρησιμοποιήσουν τα δημοσιονομικά εργαλεία του ESM στην ε, ανάκαμψη. Και προφανώς, προφανώς ε, προ, προτιμούν να έχουν χρήματα χωρίς ε, όρους και χωρίς προϋποθέσεις. Θα μπορούσαμε να έχουμε χρησιμοποιήσει το ESM ε, με τα παραδοσιακά εργαλεία, όπως είπε και ο κ. Μπρανσάρτ. Το πρόβλημα είναι ότι από τη στιγμή που κάποιες χώρες χρησιμοποιούν ε, το πρόγραμμα αυτό χωρίς ουσιαστικά όρους και προϋποθέσεις, ήταν δύσκολο να προσθεθούν αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις. Πώς λοιπόν θα τις πείσουμε να μετακινηθούν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου θυμήσατε τις καλές ημέρες που ο Ολιβιέ εργαζόταν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ήμουν αντιθύνων σύμβουλος. Πάντα εκτιμούσα τη σοφία του, το όραμά του. Είναι η πολυτέλεια ενδεχομένω του να παρατηρήσει κάτι παρά να είσαι στη μέση της διαδικασίας. Ε, εκ των υστέρων λοιπόν για το ποια θα ήταν η καλύτερη λύση αν είχαμε την πολυτέλεια της επιλογής τότε. Αλλά να σας πω με πάσα ειλικρίνεια ότι αντιμετωπίζαμε και αντιμετωπίζουμε μια παγκόσμια κρίση με λίγα προηγούμενα στην προσωπική ιστορία. Όταν συστήσαμε το πρόγραμμα κατεπήγουσας αγοράς ε, ενεργετικού για την πανδημία, θέλαμε να υποστηρίξουμε τα νοικοκυριά. Θέλουμε να επαναφέρουμε τις ε, δυνατότητες χρηματοδότησης και να επαναφέρουμε τη σταθερότητα στην αγορά που χρειαζόταν. Και το ΠΕΠ έχει τον ίδιο στόχο όπως και πολλά προγράμματα της ΕΚΤ που είναι η σταθερότητα της αγοράς. Η νομισματική λοιπόν πολιτική έχει ως σκοπό να παραμείνει σταθερότητα, να έχουμε σταθερότητα παρά του πολλαπλού κλειδονισμού. και έτσι είναι διαφορετικό εργαλείο. Αν συγκρίνουμε λοιπόν τις δύο προτάσεις, αυτή του Ολιβιέ, η οποία δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ από το ξέρετε κι εσείς, Τότε λοιπόν συζητούσαμε και βρισκόμασταν σε μια διαφορετική χώρα, όπου μια χώρα αντιμετώπιζε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Θα θυμάστε το Μάρτιο όλες οι χώρες ήταν αντιμέτωπες με δύσκολη κατάσταση. Αυτή η συμμετρική λοιπόν απειλή εξωγενής η οποία δεν ήταν ιδιαίτερα διαφορετική από χώρα σε χώρα. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα περιθώριο αμφιβολία στο μυαλό μου ότι τότε το ΠΕΠ όπως ε, δημιουργήθηκε αυτό το πρόγραμμα καταπίξεως ανάγκης ήταν η σωστή νομισματική πολιτική και έπρεπε να χρησιμοποιηθεί την περίοδο εκεί για να πετύχουμε το διτό στόχο που σας εξήγησα και προηγουμένως. Προφανώς. Όταν ε, το δημοσιονομικό και το νομισματικό σκέλος ε, συνεργάζονται όπως συνεργάστηκαν, νομίζω ότι τα αποτελέσματα και η απάντησή μας σε αυτές τις κατεπήγουσες συνθήκες είναι η βέλτιστη. Όπως ε, και εισαγωγικά αυτό το νομισματικό και το ψηλωμικό σκέλος θα πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται όσο συνεχίζει να εκτίλησεται η πανδημία χωρίς εμβόλιο μέχρι το 2021. Αλλά είναι σαφές ότι στα πλαίσια του Next Generation EU υπάρχουν δεσμεύσει και υπάρχουν συστήματα αλληλεγγύης που λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία αυτά και προφανώς θα τα παρακολουθήσετε εσείς αυτά, αυτά. Και Χαίρομαι που το ανέλαβε ως καθήκον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δούμε πού δαπανώνται οι πόροι αυτοί, γιατί θα πρέπει απαραίτητος να δαπανηθούν στους απαραίτητους ε, τομείς με τους απαραίτητους πολλαπλασιαστές για να μπορέσουμε να πετύχουμε πρόοδο. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μάρκο Τζάνι του ID έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λαγκάρτ για τη συνεισφορά σας. Δεν ακούγεται καλά ο κύριος Ζάνη. Μ' ακούτε τώρα, λέει ο κύριος Ζάνη. Είναι χαμηλός ο ήχος. I'm trying again. Can you hear me well? A bit better, but I don't think that it's enough for the interpreters, I'm, I'm afraid. Δεν είναι καλός ο ήχος, δεν έχει αρκετή ένταση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 Sorry, can you hear now me better? Loud and clear. Loud and clear. Thank you. Okay, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστούμε, ευχαριστώ κυρία Λαγκάρτ για αυτά που μας είπατε. Στην εισαγωγή σας αναφερθήκατε στον κίνδυνο και τις συνέπειες του COVID-19, της κρίσης και πολύ ψηλά επίπεδα χρέους δημοσίου και ιδιωτικού τομέα Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα αποτελέσματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο εγγύς μέλλον. Τις τελευταίες ημέρες κάποιοι και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρχίζουν να συζητούν τη δυνατότητα ακύρωσης στο μέλλον. Να ακυρωθεί, να διαγραφεί κάποιο, να ακυρωθεί ένα τμήμα των εξαγορών της ΕΚΤ. Ξέρουμε ότι υπάρχουν όρια που τίθενται στη συνθήκη. Δεν θέλω να αναφερθώ σε πολιτικές επιλογές και πολιτικές συζητήσεις. Τεχνικός πώς. Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος διαγραφής χρέους όσον αφορά την ΕΚΤ και αν οι σχετικές απώλειες από διαγραφή χρέους θα μειώσουν τη δυνατότητα της ΕΚΤ να εφαρμόσει τους στόχους της νομισματικής πολιτικής. Θα διακινδυνεύσει η χρεοκοπία η ΕΚΤ ή θα ακολουθηθούν άλλοι κανόνες από την εν συγκρίση με ιδιωτικέ τράπεζες ή άλλες εταιρείε. Μπορείτε να εξηγήσετε πως η ΕΚΤ, όπως είπε ήδη, μπορεί να εργαστεί και με αρνητικά στοιχεία ενεργητικού, αρνητικά αξιόγραφα. Είναι ειδικό ιδιαίτερο θεσμό, ειδικό θεσμό η ΕΚΤ, διαφοροποιημένο. Απάντηση, ευχαριστώ, λέει η κυρία Λαγκάρντ μου δίνει τη δυνατότητα να είμαι λακωνικότατη στην απάντησή μου. Διαβάζω με ενδιαφέρον ε, οτιδήποτε αναφέρεται, γράφεται, θίγεται, συνεντεύξεις από όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίως από αυτά, με ενδιαφέρουν αυτά που λέει ο Πρόεδρος. Απάντησή μου συντομότατη. Δεν θέτω στον εαυτό μου καν το ερώτημα. Είναι απλούστατο. Οτιδήποτε σύμφωνα με αυτά που είπατε παραβιάζει τη συνθήκη. Η ΕΚΤ λειτουργεί στα πλαίσια των συνθήκων. Υπάρχει το άρθρο 123 των συνθήκων που απαγορεύει αυτού του είδους την προσέγγιση και σέβομαι τη συνθήκη. Τελεία. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λόγο έχει. Συγγνώμη, λέει ο έχω και μπορώ να δευτερολογήσω, να υποβάλω δεύτερη ερώτηση. Έχω χρόνο. Ναι, λέει η Πρόεδρο, συγγνώμη. Συγγνώμη κύριε Τζάνι, έχετε δίκιο, έχετε χρόνο για μια δεύτερη ερώτηση. Διευκρινιστική. Mr. Zani, please go ahead. Έχετε το λόγο κύριε Τζάνι. Can you hear me now? Ακούγομαι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ξέρω ότι υπάρχουν όρια στις συνθήκες, το είπα, αλλά ίσως το μέλλον, χωρίς επίσημη διαγραφή χρέους, θα μπορούσε να έχει απόλυση η ΕΚΤ ε, λόγω των ε, στοιχείων που έχει στη διάθεσή της βάση του ΠΕΠ. Τι θα γίνει αν αυτές οι απώλειες ε, υπονομεύσουν τα στοιχεία ενεργητικού της ΕΚΤ και πώς η ΕΚΤ θα μπορούσε να ε, λειτουργήσει με αρνητική απόδοση των στοιχείων ενεργητικού της. Απάντηση. Λοιπόν, το, το σύστημα του Euro μπορεί πάντα να παράγει συμπροματική ρευστότητα ως απαιτείται. Εξορισμού λοιπόν δεν θα χρεοκοπήσει ούτε θα μείνει χωρίς χρήματα. Και πέραν αυτού, η αδίποτε οικονομική απώλεια, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, δεν θα εμποδίσει τη δυνατότητά μας να διατηρήσουμε τη σταθερότητα των τιμών και να την επιδιώξουμε. Φοβούμε ότι ξανά είναι απλούστατη η απάντηση που μπορώ να δώσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε. Δεν κάνω εικασίες επί εναλλακτικών ε, σενάριων. Έχουμε μια συνθήκη Είμαστε οι μόνοι που εκδίδουμε αυτά τα αξιογράφα και δεν ε, διατέχουμε κίνδυνο σαν αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χρόνος για άλλη διευκρινιστική ερώτηση. Νομίζω ότι όλα ήταν σαφή. Δίνω το λόγο στον Σβέν Γκίγκολτ από τους Πρασίνους. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, λέει ο κ. Έχω προβλήματα με τη σύνδεση. Με ακούτε? Σας ακούμε και σας βλέπουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Λαγκάρτ, κυρία Πρόεδρε, η ΕΚΤ αντέδρασε τολμηρά και γρήγορα και σταθεροποίησε τις ευρωπαϊκές οικονομίες στην κρίση του ευρώ και στην πανδημία. Διασταλτικά μέτρα ήταν επαρκή τα νομισματικά. Ανησυχώ για τις πρόσφατες εξελίξεις του προγράμματος του μακροπρόθεσμου επαναχρηματοδότησης, του TRTO, TLTRO. Για να προωθηθεί η δανειοδότηση από τράπεζες, τα TLTRO ευνόησαν την δυνατότητα δανειοδοτήσεων των τραπεζών. Αλλά οι στόχοι για δανειοδότηση επιχειρήσεων νοικοκυριών το 2014 επηρεάστηκαν έτσι. Με τη χαλάρωση των όρων την άνοιξη, το TLTRO 3 έγινε περισσότερο σύστημα επιδοτήσεως για τις τράπεζες της Ευρωζώνης, χωρίς αιρεσιμότητα αποτελεσματική. Αυτό οδήγησε σε με πολλά δάνεια TLTRO τον Ιούνιο. 1,3 δις ευρώ ήταν τα δάνεια. Όμως οι τράπεζες μπορούν να δανείζονται χρήματα ακόμα και πιο κάτω από το επιτόκιο καταθέσεων και με τους ρυθμούς που απορροφούν τη LTRO οι τράπεζες και τα βάζουν καταθέσεις στην ΕΚΤ είναι κερδοφόρα αυτή η κίνηση. Άρα ερώτηση. Καταρχάς, πόσες τράπεζες συμμετέχουν στο παρόν προγραμματή LTRO θα είναι επιλέξιμες για να διορτηθούν στο επιτόκιο μείον 1%. Δεύτερον, πώς εξασφαλίζεται ότι το ELTRO δίνει κίνητρα για παραγωγική δανειοδότηση που χρειάζεται για την ανάκαμψη από την πανδημία, αντί αμφισβητούμενες κινήσεις που δημιουργούν μη βιώσιμο χρέος. Τρίτον, ε, θεωρείται ότι τα προγράμματα Altiero έχουν στρεβλώσει ε, την αγορά για τραπεζικά ομόλογα. Οπότε υγιείς και μη υγιείς τράπεζες πληρώνουν παρόμοια επιτόκια για επαναχρηματοδότηση. Μπορούν οι δυνάμεις αγοράς να λειτουργήσουν ε, ακόμα σωστά όπως θα έπρεπε. Απάντηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας που αφορούν το δεύτερο κλάδο αντίδρασης ε, στην κρίση, τα Αυτό το μέσο ήταν αποτελεσματικότατο. Δύο πράγματα να πω. Το πρώτο, η επαναχρηματοδότηση, τα προγράμματα αναχρηματοδοτήσεως που δρομολογήθηκαν, δρομολογήθηκε μάλλον το πρόγραμμα με σταφή στόχο να διατηρήσει και να συνεχίσει τη δανειοδότηση εν γέννη στην οικονομία. Διότι στην αρχή της κρίσης σαφώς είδαμε ένα κίνδυνο. Κίνδυνο παγώματος της οικονομίας. Παγώματος της χρηματοδοτήσεω προ εταιρείε. Αυτό πραγματικά, αυτό ήταν ο στόχος ο επιδιωκόμενος. Σαν αποτέλεσμα αυτού πάω στο δεύτερο σημείο. Δημιουργήσαμε το πρόγραμμα αυτό αναχρηματοδότησης με βασική ερεσιμότητα. Επιτακτική ερεσιμότητα για να είναι επιλέξιμες οι τράπεζες για το ευνοϊκό επιτόκιο που αναφέρατε. Και αυτή η βασική ερεσιμότητα διατηρείται, διατηρεί τουλάχιστον τον όγκο δανειοδοτήσεως που παρήχε το πρόκρισεως COVID. Η αρχή της αιρεσιμότητας ποια είναι, ότι αν η δανειοδότηση δεν διατηρείται τουλάχιστον στο επίπεδο προ-COVID και υπάρχει σειρά ολόκληρη περίπλοκων ορίων, μετρήσεων, περιόδων αναφοράς που είμαι σίγουροι ότι γνωρίζετε και δεν θα επισέλθω εκεί αλλιώς θα, δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Αν δεν υπάρχει αυτή η αρισιμότητα, δεν, δεν πληρούνται, δεν είναι διαθέσιμο το ευνοϊκό επιτόκιο. Και πάμε στο DFR, μείον 50 σημεία βάσεως. Ο κίνδυνος αυτών των trade-offs δεν υπάρχει, δεν είναι ενταγμένος αυτός ο κίνδυνος, δεν υφίσταται στο σύστημα που δημιουργήσαμε. Γιατί ήταν επιτυχέστατο το σύστημα και χρησιμοποιήθηκε τόσο εκτενώς. Φαινομενική η χρήση του τον Ιούνιο. Γιατί, διότι καταρχάς το επιτόκιο ήταν ελκυστικό και δεύτερον οι τράπεζες θεώρησαν ότι η αιρεσιμότητα θα μπορούσε να πληρούνται και ελπίζουμε, ελπίζαμε όλοι ότι θα πληρούνται, αλλιώς δεν υπάρχει αυτό το επιτόκιο. Διότι είχαν μεγάλη ζήτηση από τι εταιρείε. Και για να ανταποκριθούν σε αυτή τη μεγάλη ζήτηση έπρεπε να χρησιμοποιήσουν και να συμμορφωθούν με τους κανόνες TLTRO. Θα είμαστε πολύ προσεκτικοί, είτε βάσει της υπηρεσίας της τραπεζών, είτε βάσει της αντιδράσεως που έχουμε από τους επιχειρηματικούς φορείς και έχουμε και έντυπα και τρόπους να αξιολογήσουμε τη βαθμολόγηση αν θέλετε και τα στοιχεία που μπορούμε να συλλέξουμε. Θα προσέξουμε ούτω ώστε το TLTRO να εξακολουθεί να κατευθύνεται προς τον σκοπό, δηλαδή συνεχή υποστήριξη της οικονομίας. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Thank ευχαριστούμε πολύ. Ρόμπερτ Ζήλε τώρα. ECR. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ, κυρία Λαγκάρτα, για την περιγραφή της μακροοικονομικής κατάστασης που μας παρουσιάσατε και για το τι πρέπει να κάνουμε και από πλευράς της δημοσιονομικής πολιτικής. Τώρα για τις λεπτομέρειες. Χτες είχαμε κάποια στοιχεία από την Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Οι διάφορες ε, χώρες αντιμετωπίσουν διαφορετική κατάσταση. Κάποιες δεν χρησιμοποιούν ε, επεκτατικά μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής. Ενώ είπατε ότι θα έπρεπε ή τις εγγυήσεις, ε, τις για τις επιχειρήσεις, για παράδειγμα. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν ότι η διάρθρωση των οικονομιών είναι διαφορετική στις διάφορες χώρες της Ευρωζώνης και τις οικονομικές προοπτικές, οι οποίες δημοσίευονται και στους Financial Times και αλλού, πότε εκτιμάτε ότι θα επιστρέψουν στο ΑΕΠ πρώτης πανδημίας οι διάφορες ε, χώρες. Γιατί από ό,τι διαβάζουμε μέχρι τώρα, άλλες θα τα καταφέρουν, άλλες δεν θα τα καταφέρουν. Και το ESM φαίνεται ότι δεν χρησιμοποιείται ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός σταθερότητα. Ούτε πολιτικά και ούτε τα δάνεια από αυτό θα χρησιμοποιηθούν. Οπότε θέλω να ρωτήσω το εξής. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να επηρεάσουμε τον δανεισμό και να επηρεάσουμε τις χώρες μέλη να χρησιμοποιήσουν επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. Πώς θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες αρχές για το πώς θα επιστρέψουμε στα ίδια επίπεδα συμφώνου σταθερότητας με τις διάφορες ρήτρε δηλαδή. Και αν δεν είναι αυτό, κάτι άλλο, ώστε να καταλάβουν οι χώρες τι πρέπει να πετύχουν μέσα στα επόμενα τρία-τέσσερα χρόνια. Θα ήταν πολύ σημαντικό. Και για τη δημοσιονομική πολιτική την επεκτατική. Επίσης, αν λάβουμε υπόψη μας τις διαφορές στις διάφορες χώρες, τα επιτόκια, εφόσον αυξηθούν, θα δημιουργήσουν ένα διαφορετικό περιβάλλον. Τώρα έχουμε το ΠΕΠ ή παρόμοια εργαλεία, αλλά τα επιτέκια είναι κάτι τα οποία θα λειτουργήσουν για όλες τις χώρες μέλη. Οπότε μήπως θα ήταν και αυτό λύση για να φέρετε σε πέρα στις αρμοδιότητές σας. Η κυρία Λαγκάρτ, ευχαριστώ πολύ για τις πολύπλευρες ερωτήσεις σας. Θα επικεντρωθώ στο παρόν. Είναι δύσκολο, έτσι κι αλλιώς, να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας σήμερα. Είναι δύσκολο να προβάλλουμε τους εαυτούς μας σε μερικά χρόνια από τώρα. Όπως λοιπόν έχει σήμερα η κατάσταση, συμφωνώ μαζί σας για το ότι είμαστε αντιμέτωποι με μια κατακαιρματισμένη κατάσταση. Και ο κατακαιρματισμός ε, αυτός έχει ως εξής. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες βασίζονται στα διάφορα προγράμματα. Παρακολουθούμε την κατάσταση. Σίγουρα είναι κάτι που μας ε, απασχολεί ε, στην ΕΚΤ και θα μιλήσουμε και γι' αυτό αργότερα σήμερα. Σε κάποιες χώρες τα προγράμματα εγγυήσεων χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς, σε άλλες χώρες όχι τόσο. Και μάλιστα για λόγους που πραγματικά δεν είναι ξεκάθαρη για μας. Υπάρχουν όμως αυτές οι διαφορές. Υπάρχει κατακαιρματισμός εξαιτία αυτού. Και παρόμοια δημοσιονομικά προγράμματα δεν χρησιμοποιήθηκαν με τον ίδιο τρόπο, είναι σαφές. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τα παρακολουθούμε αυτά. Δεύτερον, έχουμε μία εντολή για την Ευρωζώνη και παρόλο που εξετάζουμε και τις διαφορές από χώρα σε χώρα, λειτουργούμε σε επίπεδο Ευρωζώνης. Αυτή είναι η αποστολή μας. Και τρίτον, η σύνδεση της νομισματικής με τη δημοσιονομική διάσταση, όπως είπα και στην αρχή, είναι κάτι ζωτικής σημασίας οι χώρες που κάνουν προσπάθειες μεταρρυθμίσεων δεν θα πρέπει να χάσουν την ευκαιρία να προσφέρουν τα θεμέλια πάνω στο οποία η νομισματική σταθεροποίηση κατά κάποιο τρόπο και τα δημοσιονομικά μέτρα θα έχουν την ευκαιρία να μεταβάλουν τις οικονομίες τους. μπορούν να βοηθήσουν να βελτιωθεί και η παραγωγικότητα πέρα από την ψηφιακή μετάβαση κτλ. Και τα τρία αυτά θα πρέπει να πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση προκειμένου να προετοιμαστεί η Ευρώπη να είναι ένας ισχυρός παίκτη γεωπολιτικά και γεωοικονομικά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Το λόγο έχει τώρα ο επόμενος ομιλητής, αλλά να σας υπενθυμίσω, διακόπτεται πρόεδρος, α, μια στιγμή να υπενθυμίσω στους συναδέρφους. Δύο λεπτά παρακαλώ καθένας. Δημήτρης Παπαδημούλης τώρα από την ΚΟΕ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Λαγκάρτ και για την ενημέρωση που μας κάνατε. Ε, οι τελευταίες ε, εκτιμήσεις της Κομισιόν προβλέπουν μια μεγάλη αύξηση του δημόσιου χρέους ε, για όλη την Ευρωζώνη πάνω από το 100% του ΑΕΠ. Για τη χώρα μου την Ελλάδα το χρέος έχει ανέβει πάνω από το 200% του ΑΕΠ. Το σύμφωνο σταθερότητας έχει ως όριο το 60% του ΑΕΠ και οι προβλέψεις λένε ότι για αρκετά χρόνια, ίσως και δεκαετίες, θα υπάρχει μια απόκληση ανάμεσα στην πραγματικότητα και στον κανόνα. Πώς ε, βλέπετε την άποψη που υπάρχει ισχυρή μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές, αναθεώρηση σε αυτό το σύμφωνο σταθερότητας έτσι ώστε να γίνει ένα σύμφωνο σταθερότητας αλλά και βιώσιμης ανάπτυξης. Και το δεύτερο ερώτημά μου, δίπλα στην ισχυρή νομισματική πολιτική, πολλοί λένε ότι χρειάζεται και μία ισχυρή και με μεγαλύτερη διάρκεια δημοσιονομική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο με δεδομένες και τις απειλές από ορισμένα κράτη-μέλη ότι θα καθυστερήσουν ή και θα μπλοκάρουν το Ταμείο Ανάκαμψης, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς εκτιμάτε εσείς τις προτάσεις, τις σκέψεις που από ό,τι ε, ξέρω υπάρχουν και ως μελέτες και μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, που ζητούν το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει μεγαλύτερη διάρκεια από αυτήν που έχει ήδη αποφασιστεί από το Συμβούλιο και ενδεχομένως κάποια του στοιχεία να γίνουν και στοιχεία μιας μόνιμης πολιτικής δημοσιονομικής στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Σας ευχαριστώ. Η κυρία ευχαριστώ πολύ. Θέτετε σημαντικά ζητήματα. Και έχετε δίκιο ότι το COVID-19 μας οδήγησε σε ύφεση και σε μέτρα ε, στις διάφορες χώρες με αποτέλεσμα την αύξηση του δημοσίου χρέους ξέρω, είμαι σίγουρη ότι έχετε ελέγξει τα νούμερα, δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ. Και πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το χρέος έγκαιρα για να μειωθούν οι κίνδυνοι όσον αφορά το θέμα της βιωσιμότητας του χρέους και αυτό μέσω πρόθεσμα. Υπάρχουν βέβαια κίνδυνοι μιας ανάκαμψης που θα αρχίσει, οπότε βράχει πρόθεσμα χρειάζεται στήριξη από τις εθνικές δημοσιονομικές αρχές και από τη δημοσιονομική πολιτική των χωρών μελών. Κάτι το οποίο πρέπει να συνεχιστεί και οι δεσμεύσει που αναλαμβάνονται και που υπολογίζουμε και εμείς, σύμφωνα με τον προπολογισμό που υποβάλλεται, φαίνεται ότι θα συνεχιστεί η κατάσταση όπως και το 2020 σε ένα βαθμό, αλλά βέβαια όλα εξαρτώνται από το πώς θα προχωρήσει η πανδημία. Μεσοπρόθεσμοι κίνδυνοι για μη βιωσιμότητα του χρέους υπάρχουν και πρέπει να τους προσέξουμε. Θα επιστρέψουμε σε ένα βαθμό κανονικότητα βέβαια. Θα υπάρξει ανάκαμψη όπω είχαμε το Μάιο και τον Ιούνιο και ελπίζουμε πιο μακροπρόθεσμα. Κάτι το οποίο θα επηρεάσει και τον αριθμητή και τον παρονομαστή. Οπότε θα αυξηθεί το ΑΕΠ. Αλλά η βιωσιμότητα του χρέους είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ γιατί υπονομεύει την κατάσταση και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα ε, στα πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνηση. Σίγουρα, ο Πίτροπος Τζεντιλόνι ε, το έχει αναφέρει ότι θα αντιμετωπίσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έρθει με προτάσεις και οι χώρες ε, μέλη να συμφωνήσουν. Όλα αυτά βέβαια στις παραμέτρους της συνθήκης που βάζει και κάποιους περιορισμούς εννοείται. Τώρα, για το Ταμείο Ανάπτυξη και το Next Generation EU. Σίγουρα χρειάζεται καινοτομία από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και η δικιά μου ελπίδα, έτσι όπως κοιτάω εγώ τα πράγματα από τη δικιά μου προοπτική από την ΕΚΤ, είναι ότι θα εφαρμοστεί, θα αναπτυχθεί γρήγορα, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες πολλών χωρών μελών, έτσι όπως συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο και εγκρίθηκε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, κατά πόσο πρέπει να αποτελέσει ένα μόνιμο μέσο, δεν θα το αποφασίσω εγώ, ούτε μπορώ να πω εγώ τίποτα γι' αυτό. Παρατηρώ όμως ότι επηρεάζει την κατάσταση. Θα είναι αποτελεσματικό, ελπίζω, όταν θα αναπτυχθεί και μπορώ να προτείνω να εξετάσουμε το κατά πόσο ένα τέτοιο μέσο ή κάποιο αντίστοιχο μέσο με τις ίδιες αρχές να μπορούσε να επαναληφθεί σε επόμενη περίπτωση έκτακτης κατάστασης κατεξαίρεση. Τώρα πρόκειται για μια κατεξαίρεση απόφαση και ήδη είναι εντυπωσιακή σαν απόφαση αυτή που ελήφθη. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ενίκο Γκιόρη τώρα από το ΕΛΚ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και καλώ ορίσατε στη συνεδρίασή μα. Δύο ερωτήσει έχω να κάνω. Η πρώτη είναι σύντομη σε ό,τι αφορά το House. Τονίζεται διαρκώ η σημασία των πράσινων επενδύσεων. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον η ΕΚΤΕ σκοπεύει να ξεκινήσει πιο πολλέ τέτοιε στοχευμένε πράξει μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση με πράσινη ε, επικέντρωση. Δεύτερη ερώτηση, πιο δύσκολη και ακολουθώντας και την πορεία των ε, συναδέλφων. Ε, αναφερθήκατε στα προβλήματα που υπάρχουν ε, για το εξάμεινο κτλ. Στο Κοινοβούλιο αυτό το θέμα συζητιέται πολύ έντονα και πριν από κάποιες εβδομάδες εγκρίθηκε μία έκθεση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, πώς θα πρέπει να αναθεωρηθεί και για το καθεξής. Και είπατε ότι Πήγαινε καλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά μετά μας χτύπησε το COVID και ξεκίνησε η θύελα. Το δίλημα λοιπόν είναι το εξή. Για πόσο καιρό μπορούμε να είμαστε και πόσο επίκης μπορούμε να είμαστε με τη δημοσιονομική μας πολιτική. Ακολουθούνται λοιπόν χαλαρές δημοσιονομικές πολιτικές γιατί το χρειαζόμαστε κατ' για την αναζωγόνηση της οικονομίας. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Ποια είναι η βέλτιστη μίξη, το, το βελτιστό αμάγαλμα πολιτικής, ε, δημοσιονομικής πολιτικής και δημοσιονομικής πολιτικής, χωρίς να υπάρχει μόνιμη βλάβη. Και το εργαλείο ανάκαμψης βασίζεται σε δανειοδότηση. Άρα, τα βάζουμε όλα ουσιαστικά στην ε, πλάτη των ε, επόμενων γενεών. Ήμασταν λοιπόν υπέρ του εργαλείου αυτού για λόγους αλληλεγγύης καθαρά. Παρά το δεν συμφωνούσαμε, ε, θα ήθελα όμως να ακούσω την δική σας άποψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απάντηση της κυρίας Λαγκάρτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τρία αυτά βασικά ζητήματα που αναφέρατε σε ό,τι αφορά τις ε, πράσινες στοχευμένες πράξεις για μακροπροθεσμή αναχρηματοδότηση. Από ό,τι ξέρετε, έχουμε πολλές καινούργιες ιδέες, οι οποίες και εξετάζονται για το πώς μπορούμε να πρασινίσουμε ε, τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα χαρτοφυλάκια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση της στρατηγικής, να ληφθούν υπόψη και κίνδυνοι για το κλίμα ως βασικό στοιχείο. Όλοι και εγώ ιδιαίτερος προσωπικά χαίρομαι που διαπιστώνω ότι τόσοι εμπειρογνώμονες ε, σκέφτονται το κοινό καλό υπέρ του περιβάλλοντος, υπέρ της ποικιλία, ε, της βιοποικιλότητας και της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος. Καλωσορίζουμε λοιπόν όλες αυτές τις ιδέες και όλες αυτές τις προτάσεις που προκύπτουν από τις προσπάθειες που καταβάλουν. Οι διάφορες προσπάθειες οι οποίες είναι υπό εξέταση ε, διαφέρουν ω προς το πεδίο εφαρμογή το επίπεδο τεχνικών λεπτομεριών, ε, το επίπεδο υλοποίηση. Όλες οι προτάσεις έχουν κάποια αξία σε ό,τι αφορά τις πράσινες αυτές στοχευμένες πράξεις της ΕΚΤ για να προωθηθεί ακριβώς το σκέλος αυτό στις δημοσιονομικές αγορές. Αλλά όλες έχουν τους περιορισμούς του και όλες έχουν ε, αναπηλητά ζητήματα. Βασικά, το βασικό πρόβλημα είναι το τι αποτελεί πράσινο χρηματοοικονομικό προϊόν και από την άλλη να μειώσουμε το γραφειοκρατικό άχθος για όλες τις, όλους τους φορείς. Στην παρούσα φάση, παρά τις προσπάθειες όλων και του Κοινοβουλίου και με αυτό με απασχολεί ιδιαίτερος σας Ευχαριστώ ιδιαίτερος που κινηθήκατε όπως κινηθήκατε για το πράσινο αυτό κείμενο. Τμήμα εκ του οποίου έχει α, ολοκληρωθεί και ξέρω ότι συνεχίζονται οι εργασίες με το Επιτροπής και Γενικών Διευθύνσεων και χαίρομαι που από το 2022 θα αποτελεί μια πραγματικότητα αυτό το πράσινο κείμενο. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε για να οριστούν οι αποχρώσεις του μη πράσινου και να δούμε πώς θα γίνει και η μετάβαση και η χρηματοδότηση στη μεταβατική αυτή φάση. Είναι περίπλοκα τα ζητήματα αυτά. Για να μην λέμε απλά ότι έχουμε πράσινα τι, τι ε, δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια αξιόπιστη στρατηγική. Είναι πολύ σημαντικό όλες οι προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή να έχουμε τεκμήρια αξιόπιστα, γιατί θα υπάρχει προφανώς ε, αντίσταση. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι ως τμήμα της αναθεωρήσης στρατηγικής θα κοιτάξουμε όλη αυτή την γάμα ζητημάτων, τα δικά μας καθήκοντα, την εντολή μας, η οποία είναι η σταθερότητα τιμών. Προφανώς όμως όλοι θα πρέπει να επιτελέσουν το καθήκον τους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και εδώ πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ ιδιαίτερα με τον συνάδελφο από την Bundestag. Όλοι θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι «Α, δεν κάνω το καθήκον μου γιατί είναι πολύ δύσκολο». Δεν μπορούμε να περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι θα τα αναλάβει όλα. και ότι θα είμαστε ασφαλείς. Όχι. Όλοι θα πρέπει να επιτελέσουμε το καθήκον μας σε ό,τι αφορά και το πεδίο της εντολής μας. Και αυτό σίγουρα θα το προσπαθήσουμε να κοιτάξουμε όλες τις ε, δράσεις από τα πολύ καθημερινά, ε, τα κτηριακά, της οργάνωσης, μέχρι και την νομισματική πολιτική και την υλοποίηση της νομισματικής πολιτικής. Η δεύτερη ερώτηση, και πολύ φοβάμαι ότι ξεπερνά το χρόνο που μου έχει χορηγηθεί, για το ποια είναι η βέλτιστη πολιτική το βέλτιστο αμάγαλμα πολιτικών, δημοσιονομικών και νομισματικών. Κοιτώντα ε, λοιπόν την εμπειρία μου, πρέπει να σας πω ότι τα δύο αυτά πάνε χέρι-χέρι. Δεν μπαίνουμε στα χωράφια ο ένας του άλλου. Από πλευρά τη ΕΚΤ μείναμε στο πεδίο τη εντολή μας. Δεν απειλήθηκε ποτέ η ανεξαρτησία μα, ποτέ δεν μα ζητήθηκε από οποιαδήποτε δημοσιονομική αρχή να κάνουμε κάτι τέτοιο και νομίζω ότι ακριβώς τηρώντας αυστηρά τα όσα πρέπει να γίνουν στην ε, εντολή του καθενός δηλαδή, καταφέραμε να πετύχουμε αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, και καλημέρα, κυρία Λαγκάρτ. Όλοι γνωρίζουμε τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η νομισματική πολιτική στην δημιουργία θέσεων απασχόληση. Και χρειαζόμαστε λοιπόν να γνωρίζουμε ότι δεν είναι ουδέτερες οι νομισματικές πολιτικές σε ό,τι αφορά την παροχή κινητρών. Και η νομισματική και η εμπορική πολιτική σε πολλές περιπτώσεις δεν φτάνουν για να πετύχουμε το στόχο και του πληθωρισμού αλλά και την, ε, της ανεργίας, της πρόληψης της ανεργίας. Χορηγούνται όμως ε, πόροι για την ε, πρόθεση της ισότητας των φύλων και βλέπουμε ότι λαμβάνονται πρωτοβουλίες, για παράδειγμα, στην ΕΚΤ για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Ερωτώ λοιπόν, υπάρχουν ε, νομισματικά μέτρα για να προωθηθεί η ισότητα των φύλων και αν υπάρχουν τέτοιες πολιτικές. Πείτε μας μερικές πρωτοβουλίες. Αν δεν υπάρχουν όμως, η ΕΚΤ θα σκεφτεί να δράσει πιο πολύ προς την κατεύθυνση αυτή της ισότητας των φύλων η απάντηση της κυρίας Λαγκάρτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Και να πω ευθύ εξ αρχής ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως και άλλοι φορείς, έχει μία βασική εντολή και δευτερογενείς ενδεχομένως ε, εντολές. Αλλά αυτή η πρωταρχική ε, εντολή είναι η σταθερότητα των τιμών. Αυτό αποτελεί ένα ελάττωμα, θα έλεγα πως όχι. Γιατί η σταθερότητα τιμών με τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας επιτυγχάνεται με την επίτευξη σταθερότητας της οικονομίας, της γενικότερης οικονομίας. Αυτή είναι η εντολή μας, η σταθερότητα τιμών και κατά συνέπεια η σταθεροποίηση της οικονομίας. Είναι κρίσιμη αυτή η εντολή για να δημιουργηθούν θέσει απασχόληση, για να λαμβάνονται αποφάσεις, για να λειτουργήσουν αυτοί οι τομείς της οικονομίας που είναι πιο ευάλωτοι. Να έχουν πρόσβαση και αυτοί στη χρηματοδότηση. Μέσω λοιπόν της εντολής αυτής για τη σταθερότητα τιμών μπορούμε να προσπαθήσουμε να πετύχουμε το στόχο που αναφέρετε. Ένα παράδειγμα να σας δώσω. Στην παρούσα φάση είναι σαφές. Λόγω των ε, συμμετρικών αυτών και εξωγενών ε, και άνισων, αν θέλετε, κλειδονισμών, κάποιοι τομείς ε, τα πηγαίνουν καλύτερα από ότι άλλοι. Αυτοί οι τομείς έχουν να κάνουν με διπρεσίες. Κάποιοι άλλοι όμως τομείς, όπως ο τουρισμός, η ξενοδοχή κτλ. Αλλά και πιθανότατα παραδοσιακά γυναικοί τομείς Κάποιοι τομεί λοιπόν θα, θα βγουν πιο ισχυροποιημένοι μετά την κρίση. Η ΕΚΤ νομίζω παίζει το ρόλο της υπό τους περιορισμούς που έχει και βάσει της εντολής που έχει και η ΕΚΤ δίνει αυτό που χρειάζεται προκειμένου τα τμήματα της οικονομίας που υποφέρουν και κατά συνέπεια και η ανίσότητα των φύλων που υπάρχει στους τομείς αυτούς να απαλληλθεί. Δεν νομίζω ότι αρκεί αυτό από τη δική μου πλευρά, αλλά αυτό μπορεί να κάνει η νομισματική αρχή. Θα πρέπει να ληφθούν πιο πολλέ αποφάσει σε δημοσιονομικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο. Και ξέρω ότι εσείς επικεντρώνεστε στα ζητήματα αυτά και το Κοινοβούλιο ε, γενικά επικεντρώνεται σε τέτοια ζητήματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έγκυν Ερογλού από το Ρινιού. Engin Ερόγλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε και ελπίζω να με ακούτε καλά κυρία Λαγκάρτα. Σας καλωσορίζω και εγώ στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και χαίρομαι ιδιαίτερος που είσαστε τακτικά μαζί μας. Αυτό που με απασχολεί ιδιαίτερα είναι η σταθερότητα και για αντιμετώπιση κρίσεων του τραπεζικού τομέα, γιατί υπάρχει αυτή η σύνδεση μεταξύ των τραπεζών, του κράτους, της οικονομίας, πολύ απλά υπάρχει αυτή η σύνδεση. Όπω είπατε, είναι πάντα ενδιαφέρον να ακούμε τι λένε οι εμπειρογνώμονε από αυτόν. Και σε, στην ΕΦΑΤΣ, την εφημερίδα, διάβασα μία συνέντευξη του Μπουρχατ Βάλτσε από την Γερμανική Τράπεζα που ανησυχεί για το ψηφιακό ευρώ και ενδεχόμενα προβλήματα σταθερότητα του ψηφιακού ευρώ και το πώς θα επηρεάσουν τις τράπεζες. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν την δική σας άποψη. Ερωτώ, το ψηφιακό ευρώ ενδεχομένως πιστεύετε ότι μπορεί να οδηγήσει σε ένα bank run, δηλαδή ε, σε περιπτώσεις κρίσεων να φεύγουν χρήματα και να διαραίουν προς το ψηφιακό ευρώ. Αυτό θεωρώ ότι αποτελεί παράγοντα κρίσης. Είναι ένας δείκτης κρίσης. Θα ήθελα να ακούσω την δική σας άποψη από αυτό. Για το κατά πόσο το ψηφιακό ευρώ επίσης παρουσιάζει άλλους κινδύνους για μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Και πάλι θα ήθελα να πω ευθύς εξ αρχής ότι καταρχάς το ψηφιακό ευρώ όταν και αν έλθει, δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση ακόμα, δεν θα αποτελέσει υποκατάστατο των μετρητών. Θα είναι ένα συμπλήρωμα. Όχι όμως υποκατάστατο των μετρητών. Θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν λοιπόν τα νομίσματα και τα χαρτονομίσματα για όσους τα προτιμούν σε σχέση με το ψηφιακό ευρώ. Κατά δεύτερον, δεν είναι μία προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω, bottom up. Γιατί στην παράδοση του χρόνου έχουμε διαπιστώσει ότι όλοι και πιο πολλοί Ευρωπαίοι εξαρτώνται ε, και χρησιμοποιούν ε, αυτόματα συστήματα πληρωμών, ψηφιακά, ψηφιακές πληρωμές και λιγότερο τα μετρητά. Και αυτό προφανώς το επιτάχυνε η, πανδημία e-payments, ε, άμεσες πληρωμές, ε, ψηφιακές ε, κάρτες στις χώρες που δεν υπάρχουν τόσο πολλά τέτοια συστήματα αυτόματες πληρωμής. Έχει επιταχυνθεί λοιπόν η διαδικασία αυτή. Κατά τρίτον, υπάρχει ανταγωνισμός και αυτό το ξέρουμε όλοι. Υπάρχουν δίκτυα τα οποία έχουν και σημαντικές επιπτώσεις που εξετάζουν το ενδεχόμενο εισαγωγής νομισμάτων. Και αν τα λάβουμε λοιπόν αυτά υπόψη, ε, ότι δεν υπάρχει περιθώριο υποκατάστασης του νοητών ότι υπάρχει επιταχυμένη ανάγκη και ζήτηση και κατά τρίτον ότι θα πρέπει να υπάρχει θέμα κυριαρχία των Ευρωπαίων στο νόμισμά του. Γι' αυτά λοιπόν εξετάζουμε το πώς θα λειτουργούσε ένα ψηφιακό ευρώ. Αν λοιπόν είναι λιγότερο κοστοβόρο, πιο αποτελεσματικό, πιο πράσινο και να δίνει και μια καλύτερη απάντηση στη συζήτηση των πολιτών, βεβαίως. Γιατί να μην το εξετάσουμε. Για το πώς μπορούμε δηλαδή να α, περιορίσουμε την αρνητική, τις αρνητικές συνέπειες ενός ενδεχόμενου ψηφιακού ευρώ. Σίγουρα πάντως η ΕΚΤ δεν θέλει να ελαττώσει ε, και να μειώσει την νομισματική της πολιτικής και τα κανάλια της διόδους νομισματικής πολιτικής. Και πρέπει προφανώς να κοιτάξουμε πώς θα οικοδομηθεί αυτό το ψηφιακό ευρώ και σε τι σύστημα θα βασιστεί. Ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σας. Thank you. Uh, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Χωσέ Μανουέλ Γκαρίσα Γκαρσία Μαργκάιο ή Μαρσφίλ έχει το λόγο από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Έχει πρόβλημα σύνδεση ο κ. Μαργκάιο. Α πάμε στον επόμενο ομιλητή και άμα γίνει σύνδεση, επαρχόμαστε. Πάμε στον επόμενο. Γκούναρ Μπέκ από το ID. Καλημέρα, κυρία Λαγκάρντ. Να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι δεν είμαστε αντίθετοι στην αύξηση των δημοσίων δαπανών, αλλά οι περιορισμένου σκοπού όπω είναι η υγεία, η προστασία των θέσεων απασχόληση σε εθνικό επίπεδο. Σε ανταπόκριση στην επιδημία του κορονοϊού, η ΕΚΤ από το Μάρτιο αγόρασε ομόλογα και άλλα αξιόγραφα. Ήψους 870 δι ευρώ. Περίπου 7,3% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης δηλαδή. Παλιά είχαν τυπωθεί 3 εκατομμύρια, αλλά το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη συρρυκνώθηκε παρόλα αυτά με πιο οξύς ρυθμούς από ότι στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη ΣΥΠΑ, την Ιαπωνία και τον μέσο όρο του ΟΣΑ. Την περασμένη φορά σας είχα ρωτήσει αν μπορούσατε να μας δώσετε ένα απλό ιστορικό παράδειγμα που μαζική παραγωγή χρήματος οδήγησε σε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη πριν εγκαταληφθεί αυτή η πολιτική. Ερώτηση. Πόσο μεγάλο πρέπει να το ισοζύγιο της ΕΚΤ ή πόσο πρέπει να μειωθεί το ΑΕΠ της Ευρωζώνης πριν εγκαταλείψετε την πολιτική που κληρονομήσατε τον κύριο Ντράγκη. Ολοκληρώνοντας, να προσθέσω κάτι. Δεν μου αρέσει που θέτω αυτές ερωτήσεις. Ξέρω ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα πολλών πολιτικών και παραγόντων. Αλλά δεν μπορώ να σας ζητήσω να σχολιάσετε πολιτικές για τις οποίες είναι υπεύθυνοι άλλοι. Όμως, αν η Ευρωζώνη ε, αυξανόταν η παραγωγή της ε, ε, με χαμετός από τον υπόλοιπο κόσμο και η οικονομία συστέλλεται τώρα ε, με ταχύς ρυθμούς. Αυτό είναι ε, κυρίως πρόβλημα των ε, οικονομιών των, των διαφόρων χωρών και όχι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Απάντηση. Ευχαριστώ για αυτά που είπατε και τις ερωτήσεις σας, λέει η κυρία Λαγκάρτα, απαντώντας. Πρώτα απ' όλα, να αναφερθώ σε αυτό που θίξατε, τις δημόσιες δαπάνες. Τι παρατηρούμε υπό τις παρούσες περιστάσεις. ανησυχία, έλλειψη εμπιστοσύνης, τεράστια βεβαιότητα από πλευράς όλων σχεδόν των οικονομικών φορέων. Βλέποντας ε, τι γίνεται με τις επενδύσεις, με την κατανάλωση, βλέπω τα στοιχεία, τι γίνεται με τους δείκτες προσωπικής ε, κατανάλωσης, ό,τι κοιτάω, το, το είπα επανειλημμένα σε εγωικά μου σχόλια, από αυτούς που αναλύουν την όλη κατάσταση. Αβεβαιότητα είναι η λέξη κλειδί από όλα αυτά τα στοιχεία. Και είναι γεγονός ότι η παρουσία αυτής της αβεβαιότητας, οι φορείς, οι διαμορφώνονται στην πολιτική, επί των οποίων βασιζόμεθα, και από τις λίγες πηγές κάποιας βεβαιότητας οι πηγέ κάποια βεβαιότητα είναι οι δημόσιοι φορεί. Μπορεί να έχετε δική σα άποψη και ιδέε, αλλά έτσι το βλέπουμε. Και αυτό μας λένε και οι διάφορες έρευνες. Και οι βολιδοσκοπήσεις των καταναλωτών και οι βολιδοσκοπήσεις των εταιριών. Και έχουμε δει ότι όταν υπάρχουν δημόσιες επενδύσεις, και έχει αποδειχθεί ιστορικά αυτό, όταν υπάρχουν δημόσιε επενδύσει, σε εποχές μεγάλης αβεβαιότητας, προωθεί αυτή η επένδυση ιδιωτικέ επενδύσεις που είναι κάτι που απαιτείται διακαώ και ζητείται διακαώ αν θέλουμε να ξεφύγουμε από την παρούσα οικονομική κρίση. Μακροοικονομικός πώς. Δικαιολογείται απόλυτα το ότι οι δημόσιες επενδύσεις πρωτίστως να χορηγείται τώρα για να τονώσει αυτό που θα ακολουθήσει, δηλαδή ιδιωτικές επενδύσεις και επαναφορά της εμπιστοσύνης για τους οικονομικούς φορείς. Τι βλέπω εγώ, τι παρατηρώ βάσει των όσων κάναμε. Το μέγεθος του προγράμματός μας του κατεπήγοντος για την πανδημία. Η μεγάλη απορρόφηση των TLTROs και τα αποτελέσματα που παρήχθησαν βλέποντας όλους τους δείκτες, όγκος δανειοδότησης, επιτόκια δανειοδότησης, σταθερότητα χρηματοπιστωτικών αγορών, όροι χρηματοδοτήσεως εν γέννη. Όλα αυτά ακολουθούν μία κατεύθυνση, την κατεύθυνση της υποστήριξης των πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει. Και δεν νομίζω ότι υπήρξε εναλλακτική και ότι υπάρχει εναλλακτική υπό τις παρούσες περιστάσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν ο κύριος Γκαρσία Μαργκάγιο έχει συνδεθεί τώρα. Όχι ακόμα κυρία Πρόεδρε, προσπαθεί. Πάμε στον επόμενο μιλητή πρώτα. Μάλιστα. Γιακίμ Σούστερ ε, του, ε, των συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Νόμιζα ότι θα καθυστερούσαμε λίγο. Όπως ακούσαμε, ως τώρα στην κρίση υπήρχε καλή, καλός συγκερασμός νομισματικής ε, και δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτό δεν ήταν πάντα έτσι πριν την κρίση, αλλά ήδη υπάρχουν ε, κάποια προβλήματα πάλι και σε διάφορες περιπτώσεις ε, γίνεται απόπειρα για εγωιστικούς, εθνικιστικούς λόγους, εθνικούς λόγους να μπλοκάρουν τον ε, προπολογισμό. σε μια νομισματική πολιτική με νομισματική πολιτική κοινή, αλλά ξεχωριστή τη μεσονομική πολιτική, παρουσιάζονται λοιπόν τέτοια προβλήματα. Τώρα λοιπόν επικεντρωνόμαστε τι θα κάνουμε μετά την τρέχουσα κρίση. Θα πρέπει να μειώσουμε πάλι το χρέος και σε τι χρονικό διάστημα, τι θα γίνει με τα επιτόκια που είναι πολύ χαμηλά στην παρούσα φάση ε, και ευνοούν ε, προφανώς τις επενδύσεις, αλλά έχουν αρνητικές επιπτώσεις διαφορετικές. Πώς αναμένουμε να εξελιχθεί και ο πληθωρισμός. Σε όλες αυτές τις ερωτήσεις, καλό θα ήταν υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Άρα, ρωτώ λοιπόν κυρία Λαγκάρντα, εσείς ε, τι, ε, πώς θα συνδράμετε σε αυτό την συνδυασμό νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εμπειρίες της κρίσης για να κάνουμε θεσμικές αλλαγές και αν ναι, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνει βασικά εσείς από πλευρά σας. Uh, Ευχαριστώ πολύ για το πλαίσιο που θέσατε και τις ερωτήσεις. Συμφωνώ απολύτως. Στην παρούσα κρίση είδαμε αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ δημοσιονομικών πολιτικών και νομισματικών. Πιστεύω και διατείνομαι ότι δεν κυριάρχησε η δημοσιονομική επί της νομισματικής και η νομισματική πολιτική διατήρησε την κυριαρχία της και η ΕΚΤ παρέμεινε εντελώς ανεξάρτητη. Δεν διατείνομαι ότι είναι ο τέλειος συνδυασμός, αλλά ήταν αποτελεσματικότατος. Μ' αρέσει να δίνω παραδείγματα και δεν έδωσα μου κανένα παράδειγμα της συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ δημοσιονομικού και νομισματικού. Δεν ήταν ε, από πρόθεση. Οι αρχές το αποφάσισαν. Αναγκαία χρηματοδότηση οικονομίας ήταν ο παράγων. Από τη μία μεριά, από την αρχή, 18 Ιουνίου, δημιουργήσαμε ελκυστικότατες επιχειρήσεις αναχρηματοδότησης μακροχρόνιας, δεν θα έλεγα θαυμάσια, πώς να το πω, άλλο όρο χρησιμοποιήσω, σημαντική απορρόφηση αυτό το μέτρο, αυτό το σύστημα. Απ' την άλλη, οι δημοσιονομικές αρχές αποφάσισαν αντίστοιχα σε εθνικό επίπεδο και μετά σε ευρωπαϊκό επίπεδο να θέσουν συστήματα εγγυήσεων άνευ των οποίων οι τράπεζες πιθανότατα θα ήταν πολύ πιο διστακτικές να δανειοδοτήσουν τις εταιρείε, τους εμπορικούς φορείς, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, του επιχειρηματίες. Οπότε έχετε το παράδειγμα ζήτησης χρηματοδότηση που ήταν διαθέσιμη και τα συστήματα εγγυήσεων που θεσπίστηκαν σε εθνικό και συμπληρώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όταν αυτό χρειαζόταν. κάτι που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί απόλυτα για να συμπληρωθούν οι εγγύησει. Ένα τυπικό παράδειγμα που η νομισματική, η δημοσιονομική πολιτική χέρι με χέρι ανταποκρίθηκαν σε μια ανάγκη που ήταν κρίσιμη σημασία για να στηριχθεί η ανάκαμψη και να βοηθηθεί η οικονομία. Όπως παρατηρήσατε, τα επιτόκια, ένα τμήμα Τη παραδοσιακή εργαλειοθήκης κεντρικής τράπεζα είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Και έχουμε και κάποιες κατευθύνσει που δίνονται στην εργαλειοθήκη που δείχνουν εάν και πότε θα αλλάξουν τα επιτόκια. Και ξέρετε, αν το παρατηρήσετε αυτό και δείτε τι λένε οι σχολιαστές για το χρονισμό, το θέμα ξαφνική αλλαγή των επιτοκίων, αυξήσεω των επιτοκίων δεν θα πρέπει να είναι κάτι που να ανησυχεί εσά που ενδιαφέρεστε τα επιτόκια για τα χρέη, για το χρέος. Ήδη είπα ότι ο όγκο του χρέους και τα ποσοστά που χρησιμοποιούνται, τα, τα κλάσματα που χρησιμοποιούνται ε, χρέος έναντι ΑΕΠ δείχνουν την κατάσταση ποια είναι. Και για να κατευθύνουμε την ανάπτυξη, για να αυξήσουμε βιώσιμα το ΑΕΠ, αυτή έχει σαν στόχο να μειώσει αυτό το λόγο ε, ΑΕΠ προς χρέος. Νομίζω άλλος τομέας όπου οι δημοσιονομικές αρχές έπαιξαν το ρόλο τους για να βοηθήσουν την νομισματική πολιτική να παίξει το ρόλο της και να στηρίξει την οικονομία ήταν όταν χρησιμοποίησε ισχύοντα εργαλεία στο Σύμφωνο Σταθερότητας και ανάπτυξη, όπως η ρήτρα διαφυγή που πραγματικά ήρθε αρκετά έγκαιρα, ούτω ώστε να ενθαρρυνθούν οι εθνικές αρχές να κάνουν τα δέοντα. Και οι όροι για κρατικές ενισχύσεις ήρθαν επίσης για να βοηθηθεί η στήριξη κάποιων ιδιαίτερα ε, πληγέντων τομέων. Όλα τα χαρακτηριστικά των μέτρων πρέπει να αναλυθούν. Αυτά θα αναθεωρηθούν τα μέτρα και τα πακέτα αυτά των μέτρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα γίνει μια ισβάθωση συζήτηση για τα θέματα για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Υπάρχουν εργαλεία, αυτή είναι η παρατήρησή μου, που ήταν χρήσιμα εργαλεία και εξυπηρέτησαν τις παρούσες περιστάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ενρίκε Χαν από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ που είστε εδώ, κυρία Λαγκάρντ. Ο COVID-19 τράβηξε την προσοχή του κοινού από τους κινδύνους του κλίματος που αντιμετωπίζουμε σήμερα και αύριο και τις πυρκαγιές, τους κυκλώνες και τις πλημμύρες που οδήγησαν σε απώλειες ζωών, ανθρώπων και ζωών και επηρέασαν πολύ αρνητικά και την οικονομία και την οικονομική σταθερότητα οι τράπεζες μέσω κοινωνικής ευθύνης ε, ε, αντιμετώπισαν το θέμα. Οι αλλαγές του κλίματος πρέπει να υπολογιστούν κατάλληλα στη δημοσιονομική ανάλυση και διαχείριση κινδύνου των τραπεζών. Η Τράπεζα Διεθνών Διευθετήσεων ε, δημοσίευσε έκθεση. Συμπεριλαμβάνει άποψη όρων συμπεριλαμβανομένων ΕΚΤ για πρωτοβουλίε για κινδύνου που δημιουργούνται από αλλαγή του κλίματο. Πολλοί σημείωσαν ότι τώρα δεν υπάρχει ρητή εντολή που έχει ανατεθεί για αυτό το θέμα. Είπαν όμω ότι οι κίνδυνοι μπορεί να έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην ασφάλεια τραπεζών και ίσως δημιουργήσουν προβλήματα ευστάθεια για το δημοσιονομικό σύστημα, το χρηματοστικό σύστημα. Μέχρι τώρα η ΕΚΤ εστιάστηκε επιβεστητοποίησεω και προσανατολισμών. Η ΕΚΤ όμω δεν εφάρμοσε αποτελεσματική εποπτική προσέγγιση της τράπεζας σχετικά με τον κίνδυνο από το κλίμα, την αλλαγή του κλίματος. Δεν μας στάνει να αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα της αλλαγής του κλίματος, αντιμετωπίζουμε και με αυτά τα προβλήματα. Τα οικονομικά. Τι οδικό χάρτη έχετε για εφαρμοστικά μέτρα συμπεριλαμβάνονται και κίνδυνοι από το κλίμα στον εποπτικό μηχανισμό και να εξασφαλίζουν σαφέστατα το ότι οι τράπεζε θα χειρίζονται τον κίνδυνο του κλίματο σωστά για να αυξηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα Ευχαριστώ πολύ. Απάντηση. Διακοπή της σύνδεσης με την κυρία Λεγκάρτ. Είναι θέμα εποπτικό. Α, α, α, είμαι, είμαι, εντάξει, είμαι στην οθόνη. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Κοιτάξτε, σκεφτόμουν το εξή, ότι ένα μέλο του ερωτήματό σα αφορά υποπτικέ δραστηριότητε της ΕΚΤ. Ο Ανδρέα Ενρία ε, θα αναφερθεί σε αυτό το θέμα στην ΕΚΟΝ. Εγώ ανησυχώ. Έχω υπόψη αυτά τα προβλήματα του κλίματος. Θέλουμε να καλύψουμε όλους τους τομείς αρμοδιότητας της εντολής μας. Ξέρω ότι το υποπτικό σύστημα υποπτήρες τραπεζών έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθούν οι τράπεζες. Ο φορέας μάλλον διαχείριση του κινδύνου έχει εντοπίσει κατευθύνσεις γραμμές για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι από το κλίμα και να μπορούν να ενημερώνουν τους κινδύνους. Από ό,τι θυμάμαι, αυτό είναι κάτι που πρέπει να ενεργοποιηθεί το 2022, ούτως ώστε οι τράπεζες να ενημερώνουν περί των κινδύνων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως ξέρετε, είναι μέλος του NGFS, NGSFS, που είναι το δίκτυο για πράσινη χρηματοδότηση και συμμετέχει ενεργά στο δίκτυο. Ιδιαίτερα χαίρομαι που ο παρόν πρόεδρος του NGFS, ο Φρανκ Έντελσον, έτυχε τις εγκρίσεώς σας όσον αφορά την υποψηφιότητα για να γίνει μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα και χαίρομαι που θα φέρει τις γνώσεις του και το πάθος του για αυτά τα θέματα. Εκεί συμπεριλαμβάνω τη βεπικιλότητα. Πιστεύω ότι συμφωνείτε κι εσείς. Εν κατακλείδη. Ο υποπτικός κλάδος της ΕΚΤ λαμβάνει σοβαρότατα υπόψη αυτά τα θέματα. Το σύστημα ελέγχεται όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων. Πρέπει να αναφέρονται αυτοί οι κίνδυνοι, πρέπει να αναλύονται αυτοί οι κίνδυνοι από πλευρά τραπεζών και των τραπεζικών συστημάτων υπό του, που ελέγχονται το σύστημα ελέγχου των κινδύνων. Και σαν ΕΚΤ εμείς θα εξετάσουμε όλα τα θέματα, όλα τα χαρτοφυλάκια, το δικό μας χαρτοφυλάκιο, και εκείνα που έχουμε στη νομισματική μας πολιτική για να δούμε πώς μπορούμε τον καλύτερο τρόπο να πετύχουμε τα σωστά αποτελέσματα σύμφωνα με την εντολή μας. Χωρίς να καθορίζουμε εμείς ποια είναι η σωστή τιμολόγηση και αποτίμηση. Αυτό δεν είναι κάτι που εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Σχετικής Τράπεζας. Αυτοί που διαμορφώνουν την πολιτική έχουν τη δικαιοδοσία. Στο νομοθετικό και εκτελεστικό κλάδο να κινηθούν κατάλληλα και να ενεργοποιήσουν τους φορείς του ιδιωτικού τομέα και το IFRS Φερρυπίν για να εντοπιστούν σωστά τα προβλήματα, να καταγραφούν οι κίνδυνοι, ούτως ώστε να γίνει σωστή τιμολόγηση. Προς αυτές τις κατευθύνσεις λοιπόν πρέπει να κινηθούμε, λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή του κινδύνου και την αλλαγή του κλίματος και τους κινδύνους που συνεπάγεται και τις εξελίξεις όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος να λαμβάνονται αυτά υπόψη, ούτω ώστε να μπορούμε να, να προσμετρήσουμε τη σταθερότητα των τιμών και του σχετικούς στόχους, ένα παράδειγμα. Πώς καθορίζουμε τον πληθωρισμό, πώς προβλέπουμε τον πληθωρισμό, αν έχουμε μαζική επανάληψη καταστροφικών ε, καιρικών φαινομένων, πώς θα προσμετρήσουμε τον πληθωρισμό, αν ένας φόρος άνθρακα εφαρμοστεί στο σωστό επίπεδο τελικά. Αυτές οι δύο συνιστώσεις έχουν άμεση ή έμεση επίδραση στον πληθωρισμό. Και αυτό έχει τεράστια σημασία για την εντολή μας για τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Δύο παραδείγματα από την εποπτική πλευρά διαχείριση των κινδύνων και από την νομισματική πολιτική από την άλλη και τους στόχους. Και για τους δύο αυτούς στόχους έχει σημασία η αλλαγή του κλίματος. Uh, very Σας ευχαριστούμε πολύ. Στο μεταξύ, ο κύριος Γκαρθία Μαργάγιο κατάφερε να ξεπεράσει τα προβλήματα που είχε για σύνδεση και τώρα του δίνω το λόγο για την ερώτησή του. Κύριε Μαργάγιο, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ομιλία, παρακαλώ. A ver. Mr. Magallo, we could briefly... hear... Κύριε Μαργάγιο, ξανά το κουμπί ομιλία παρακαλώ. Okay, uh, Η Πρόεδρος. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε όσο προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα ο κύριος Καρθία Μαγκάγιο, περνάμε στην ε, Αγνές Ευρέν. ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που έχουμε την Κριστίν Λαγκάρτ ε, μαζί μας. Την ευχαριστώ λοιπόν που ήρθε. Η πανδημία COVID-19 και η κανόνες αποστασιοποίησης έχουν αλλάξει τον τρόπο της ζωής μας, τον τρόπο πληρωμών. Από τον Μάρτιο διαπιστώνουμε ότι πολύ περισσότερες συναλλαγές γίνονται ανέπαφα, αλλά μία πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι κάποιοι από τους πολίτες μας ανησυχούν για την ασφάλεια αυτού του είδους πληρωμής. Οπότε, κυρία Λαγκάρντα, θέλω να ρωτήσω δεδομένου ότι υπάρχουν κίνδυνοι για πάτες ε, ε, στον κυβέρνο χώρο κτλ. Δεν πιστεύετε κι εσείς ότι πρόκειται για απειλή στην νομισματική σταθερότητα και ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να δημοσιεύσει μια μελέτη όσον αφορά τη συμπεριφορά πληρωμής των καταναλωτών, εσείς τι μαθήματα θα πάρετε από αυτή τη μελέτη και πώς βλέπετε την αναγκαιότητα να συνδυάσετε ε, την ψηφιακή διάσταση με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών προκειμένου να επιτυγχάνεται η νομισματική σταθερότητα πάντα. Η κυρία Λαγκάρτ, ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Και εγώ χαίρομαι που σας άκουσα. Λοιπόν, τι κάναμε. αρχές Οκτωβρίου, 8 ή 10 δεν θυμάμαι ακριβώς, εκδώσαμε ένα έγγραφο ε, στο οποίο αναλύονται τα χαρακτηριστικά ενός ε, λιανικής χρήσης ψηφιακού ευρώ και εντοπίσαμε τα ωφέλη, τους κινδύνους, ε, τα θετικά αρνητικά και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Και μετά ξεκίνησε η διαβούλευση, η οποία ξεκίνησε στα μέσα Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιανουαρίου. Οπότε προς το παρόν δεν έχω αποτελέσματα από την διαβούλευση αυτή για να σας πω κάτι. Ειλικρινά δεν γνωρίζω τι υπάρχει. Ξέρω ότι έχουν συμμετάσχει πολλοί, οι συνήθεις ύποπτοι βέβαια, αλλά όχι μόνο και πολλοί άνθρωποι από το κοινό που εκφράζουν την απόψή τους απλώς. Και εννοείται ότι θα τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη όταν θα προχωρήσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο για να προτείνουμε ένα σχέδιο. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι πέρα από τις ανησυχίες της νομισματικής πολιτικής, τα θέματα της μετακύλης νομισματικής πολιτικής, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Όπως είπατε, υπάρχει και το θέμα της ασφάλειας. Ο κίνδυνος δηλαδή διείσδυσης κάποιου απ' έξω, αλλά υπάρχει και ο κίνδυνος οι ιδιωτικές πληροφορίες να διασφαλίζονται, να παραμένουν ιδιωτικές και άρα να προστατεύονται οι ψηφιακές συναλλαγές ως προς αυτό. Αυτό φυσικά και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Αλλά ακριβώ επειδή υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πέρα από τις τεχνολογικές επιλογές στις οποίες θα προβούμε, δεν είναι ένα σχέδιο το οποίο σε έξι μήνες ή ένα χρόνο θα έχει υλοποιηθεί. Σίγουρα θα χρειαστεί περισσότερο και θα χρειαστούν και περισσότερες διαβουλεύσεις. Στο μεταξύ πάντως αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό την ονομασία ΜΙΚΑ. Σίγουρα θα τη γνωρίζετε. Γιατί υπάρχει αρχή ότι η ίδια δραστηριότητα, οι ίδιοι κανόνες, αυτή η αρχή πρέπει να εφαρμοστεί. Και όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν νέοι που μπαίνουν στην αγορά και θα πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες, την ίδια εποπτεία και να λογοδοτούν με τον ίδιο τρόπο σε πολύ υψηλέ προδιαγραφέ και για την προστασία του ιδιωτικού βίου και για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων και οποιοδήποτε άλλου δεδομένου. Οπότε είναι διτή απάντησή μου. Αυτό που κάνουμε θα διέπεται από διαφάνεια. Και από την άλλη αυτό που λέτε εσείς για την προστασία της σταθερότητας του ιδιωτικού βίου και της ασφάλειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει τώρα ο Τζιν Γιουρτζίκα. ECR. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λαγκάρτ, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αρχίσει να αγοράζει πράσινο ομόλογα και να τα δέχεται σαν εξασφάλιση από τις αρχές της επόμενης χρονιάς. Θα ήθελα εδώ να εκφράσω τις ανησυχίες μου, γιατί τα πράσινα ομόλογα ενδεχομένως να παραβιάζουν την κύρια εντολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είναι η σταθερότητα τιμών. Συνεπώς θα έπρεπε η νομισματική πολιτική να είναι ανεξάρτητη και ουδέτερη όσο γίνεται περισσότερο. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αγοράζοντας ε, ομόλογα μιας εταιρεία που το ονομάζει πράσινα, παραβιάζει αυτήν την αρχή. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής λοιπόν και του περιβάλλοντος, πώς το βλέπετε ως μέρος της εντολής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και έπειτα στο μέλλον θα μπορούσε, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αρχίζει να αγοράζει ομόλογα φαρμακευτικών εταιριών με το επιχείρημα ότι η δημόσια υγεία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λαγκάρτ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Πρώτα απ' όλα, ήδη αγοράζουμε πράσινα ομόλογα. είναι μέρος των προγραμμάτων αγοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία αγοράζει, θα μπορούσα να ελέγξω τα νούμερα για να σας τα επιβεβαιώσω, αλλά εν πάση περιπτώσει περίπου 20% των διαθέσιμων πράσινων ομολόγων αγοράζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και περιμένουμε περισσότερες εκδόσεις πράσινων ομολόγων από διάφορα σημεία της Ευρώπης. Οπότε αυτή η τάση ε, αγοράς δεν θα μειωθεί. Ήδη λοιπόν αγοράζουμε πράσινα ομόλογα, ήδη τα δεχόμαστε ως ε, εγγύσεις, ως εξασφαλίσεις. Αλλά νομίζω ότι αυτό στο οποίο αναφέρεστε εσείς είναι η απόφαση που ελήφθη να δεχτούμε εξαίρεση όσον αφορά την δομή των πράσινων ομολόγων που δεχόμαστε που έχει σαν αποτέλεσμα ένα μεταβλητό το κομερίδιο αντί για σταθερό όπως ήταν πριν. Κάτι το οποίο βοηθάει να δεχτούμε ως εξασφαλίσεις κάποια από αυτά τα πράσινα ομόλογα που έχουν σχέση με το κλίμα και διέπονται από κάποια βεβαιότητα. Οπότε αυτό είναι που θα αρχίσει να ισχύει από 1η Ιανουαρίου αλλά αναφέρεστε και σε ένα γενικότερο ζήτημα βέβαια, το οποίο έχει να κάνει με τον ρόλο της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοπικιλότητας μέσω της νομισματικής μας πολιτικής. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί πάρα πολύ στο Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια της επανεξέτασης της στρατηγικής μας διότι πρέπει να εξετάσουμε την εντολή μας και σύμφωνα με τις προβλέψεις, τις διατάξεις των συνθήκων που λένε ότι η κυρία εντολή μας είναι σταθερότητα τιμών με ε, δευτερεύοντες στόχους που αναφέρονται επίσης, η προστασία των αρχών της ελεύθερης αγοράς, πρέπει δηλαδή να στηρίζονται με τις κατάλληλες πληροφορίες και τον ε, ισολογισμό κινδύνων. Οπότε, δύο πράγματα. Όταν πρόκειται για τη μέτρηση της σταθερότητας τιμών, όπως είπα και νωρίτερα, το θέμα της ε, άμεσης ή έμεσης κλιματικής αλλαγής σίγουρα παίζει ρόλο. Το δεύτερο, τι εργαλεία διαθέτουμε και τι περιθώριο ελιγμών διαθέτουμε για τον καθορισμό του πληθωρισμού. Εδώ πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τα εθνικά επιτόκια μειώνονται, μπορεί να μειώνονται ακόμα περισσότερο. Αν δούμε περισσότερες αποτομιεύσεις από τους καταναλωτές και αυτό επηρεάζει τα πράγματα. Φοβούνται λόγω της πανδημίας και αποτομιεύουν περισσότερο. Οπότε στην αξιολόγησή μας θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Συνεπώς, επηρεάζει άμεσα η κλιματική αλλαγή, το πώς μετράμε το στόχο της σταθερότητας τιμών και τι κάνουμε γι' αυτόν. Τώρα πώς αυτό με τη σειρά του επηρεάζει την νομισματική μας ε, πολιτική και τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων μας, αυτό καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι δικό του καθήκον, βάσει των όσων ανέφερα, δηλαδή βάσει των όσων αναφέρονται στις συνθήκες. Και λαμβάνοντας υπόψη την τήρηση των αρχών της αγοράς. Οπότε πρέπει να δούμε κατά πόσο η κίνδυνη, η διαφάνεια είναι πράγματα τα οποία θα επηρεάσουν το τι θα κάνουμε τελικά με τις εξασφαλίσεις και με τις αγορές ενεργητικού. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ας προσπαθήσουμε για μια ακόμα φορά να έχουμε τον κύριο Γκαρσία Μαργάγιο. Για να δούμε. Α, με βλέπετε τώρα, με ακούτε. Ναι, κύριε Μαργάγιο. Ωραία. Ευτυχώ επιτέλους, λέει ο κύριος Μαργάγιο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να κάνω μία δήλωση και μετά μία διαπίστωση και τρίτον να σας παρουσιάσω ένα πρόβλημα. Η δήλωσή μου είναι ότι δεν υπάρχουν λογικές αναλλακτικές στα μέτρα τα οποία έχουν εγκριθεί μέχρι τώρα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τα επιτόκια, τη ρευστότητα, την αγορά ενεργητικού, ε, πρόγραμμα το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό και ανταποκρίνει τις ανάγκες. Από πλευρά της ε, Επιτροπής επίσης ευελιξία των κανόνων του Συμφώνου σταθερότητα και στο Συμβούλιο σχέδιο ανάκαμψη, το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή όσο γίνεται πιο γρήγορα. Τώρα, η διαπίστωσή μου είναι ότι οι χώρες μέλη, χάρη στην ευελιξία της Επιτροπής και στη δράση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μπορεί να προσφέρει χρηματοδότηση κάτω από ικανοποιητικές συνθήκες. Ε, δίνεται ευελιξία και σε χώρες που έχουν αρκετά περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας, αλλά και στις χώρες που έχουν λιγότερα περιθώρια. Οπότε, από πλευράς καθαρά πολιτικής, ε, πολιτικού ορθολογισμού. Είναι λογικό οι χώρες που έχουν λιγότερο περιθώριο να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στην αγορά ή πρέπει να συμμορφώνονται προς το ε, προς τα όσα έχουν συμφωνηθεί μέχρι τώρα. Οπότε θέλω να ρωτήσω ότι στο βαθμό που αυξάνεται το χρέος. Οι αγορές θα αρχίσουν να κάνουν κάποια διάκριση, θα δίνουν προτεραιότητες στις χώρες ανάλογα με το μέγεθος του χρέους τους και της αξιοπιστίας τους. Οπότε πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στο πού πάνε τα χρήματα τα οποία φτάνουν από κάποια πηγή χρηματοδότησης. Να δαπανώνται δηλαδή με το σωστό τρόπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επειδή η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας είναι και επικεφαλής του Συμβουλίου Συστηματικού Κινδύνου, αυτό πρέπει να το έχει υπόψη της, γιατί κάποια στιγμή θα δημιουργηθεί αυτή η διάκριση από τις αγορές που θα διαφοροποιήσει και θα ενισχύσει τις διαφορές μεταξύ των χωρών. Έχω δίκιο ή όχι. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ. Η κυρία Λαγκάρτ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Μου δίνετε έτσι την ευκαιρία να πω μερικά πράγματα και το ένα είναι ότι δεν είμαι σίγουρη ότι πολιτική και ορθολογισμός πάνε μαζί. Δεν έχω συναντήσει πολύ πολιτικό ορθολογισμό στην ε, σύντομη αλλά έντονη ε, θητεία μου. Θέλω όμως να υπογραμμίσω ότι ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, κυρίως με το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς ενεργητικού λόγω πανδημίας, το ΠΕΠ, ήταν αποτελεσματικό, γρήγορο και ανταποκρίθηκε στην, στο διτό του σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Συνεπώς ήταν και παραμένει ένα μέσο νομισματικής πολιτικής. Δεν συνδέεται με κάποιο είδους αιρεσιμότητα. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Οπότε δεν μπορώ να σας πω ότι σκέφτονται οι αγορές, δεν είμαι οι αγορές. Είμαστε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες προκειμένου να φέρουμε σε πέρα στην εντολή μας. Ευχαριστώ. Κύριε Μαργκάια, αν θέλετε, έχετε λίγη ώρα για να κάνετε μία ερώτηση. Ιδάλλως μπορούμε να περάσουμε και στη συνέχεια. Μάλιστα, πολύ ωραία. Δεν ζητάτε το λόγο για επερώτηση. Μου είχε ζητηθεί το Catch the Eye. Δεν μπορώ να δώσω το λόγο σε μη γιατί αυτό έχει οριστεί από τους συντονιστές για το Catch the Eye. Θα δώσω λοιπόν στο λόγο στον κύριο Λευτέρη Νικολάου και στον Άλβαρο. Αλλά ένα λεπτό μόνο γιατί δεν έχουμε χρόνο, παρακαλώ. Mr. Alavanos, are you connected? Κύριε Νικολάου Αλαβάνο,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 Υπάρχει πρόβλημα τη σύνδεση το κ. Ζητώ συγγνώμη. Αλλά έχουμε ξεπεράσει το χρόνο που προβλεπόταν κατά 11 λεπτά. Ίσως να περάσουμε στην επόμενη ακρόαση. Και θα μπορούσε ίσως να ζητήσει το λόγο στο τέλος της επόμενης ακρόασης που είναι και πάλι με την κυρία Δαγκάρτα. I have uh, the Connection is uh, reinstated. Yes, please go ahead. Just one minute, please. Ναι, ναι, για ένα λεπτό παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, I ε, Greek. Πολλέ φορέ έχουμε συζητήσει σε σχέση με τα προνομιακά και δανεισμού τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προ Εθνικέ Τράπεζε για την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών, την ανάγκη για Τραπεζική Ένωση, τι απαιτήσει δηλαδή των μονοπωλιακών ομίλων για να συνεχίζουν να κερδοφορούν όπω έχετε υπεγραμμίσει, αυτό που διατράσσει το σχέδιο, μεταξύ άλλων, είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και δίδεται γραμμή και με το χθεσινό δελτίο τύπου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σε τράπεζε, funds, κυβερνήσει να πάρουν μέτρα με χιλιάδε πληστηριασμού κατοικιών, κατασχέσει λογαριασμών οικογενειών που ζουν στα όρια τη εξαθλίωση. Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση έφερε νέο νόμο για το λεγόμενο πτωχευτικό κώδικα, με τι ευλογίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση αυτόν, τελειώνει η τυπική προστασία τη πρώτη κατοικία, καθιερώνεται για πρώτη φορά πτώχευση φυσικού προσώπου ακόμη και για 30.000 ευρώ για καθυστερήσει ακόμη και 6 μηνών. Τη στιγμή που φουντώνει η ανεργία, οι απολύσει, χωρί αποζημίωση, χιλιάδε άνθρωποι βρίσκονται χωρί καν επίδομα ανεργία. Το σύνολο τη περιουσία, η κόπη μια ζωή, θα πάνε στα χέρια των πιστωτών, στα αρπακτικά τραπεζών και φαντ, για την αποπληρωμή χρεών. Ολόκληρε οικογένειε δηλαδή καλούνται να επιβιώσουν με τι λεγόμενε εύλογε δαπάνε διαβίωση 600 ευρώ, ενώ αντιμετωπίζουν και πιθανέ ποινέ φυλάκιση. Η ερώτησή μου είναι εξή. Πώ τοποθετήσετε στο αίτημα για απαγόρευση πληστηριασμών λαϊκή κατοικία και δέσμευση λογαριασμών από τράπεζε και ιδιωτικά funds. Πώ τοποθετήσετε για τη δραστική μείωση των, την απέτηση για δραστική μείωση των χρεών των λαϊκών οικογενειών στι τράπεζε, διαγραφή τόκων, ουσιαστικό κούρεμ χρέου, ώστε να δοθεί πραγματική διέξοδο και όχι παρατεταμένη ομοιρία εργαζομένων και βιοπαλαιστών αυτοαπασχολούμενων. Ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστώ. Και καταρχάς να πω ότι ε, εγώ προσωπικά συμπάσχω, συμπάσχω πολύ με όσους ε, πάσχουν. Είναι οι πιο ευάλωτοι οι γυναίκες, ε, τα χαμηλά εισοδήματα, τα παιδιά. Αλλά από πλευρά της ΕΚΤ, από τη θέση μου, δεν υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Αυτό προφανώς ε, θα πρέπει να επιληθεί σε άλλο επίπεδο και όχι στο δικό μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Λέει πρόεδρος. Και τώρα, έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη ακρόαση, ο διάλογος. Να περάσουμε στην επόμενη ακρόαση με την πρόεδρο Λαγκάτ ως πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου αυτή τη φορά. Είναι η δεύτερη φορά λοιπόν που έχει εμφανιστεί στην ΕΚΟΝ υπό την ιδιότητά της αυτή σε ό,τι αφορά το ρόλο της ε, και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου που έχουν μεγάλη σημασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προφανώ είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μα. Όπω τα ξέρουν οι βουλευτέ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, συνεχίζει τη δουλειά του για του κινδύνου που προκύπτουν από την πανδημία και έχει κάνει και σχετικέ παρεμβάσει ω προ αυτό. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν την ίδια πρακτική. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Λαγκάρτ για 15 λεπτά και στη συνέχεια θα ακολουθήσει γύρω έρτα απαντήσεων. Έχετε το λόγο, κυρία Λαγκάρτ. Μπορώ να σας ζητήσω δύο λεπτά, παρακαλώ, να πάω στην τουαλέτα. Βεβαίως, λέει ο Πρόεδρος. Βεβαίως, βεβαίως. Διακόπτουμε ασφαλώς για λίγο. Διακόπτουμε για λίγο και θα επανέλθουμε σε λίγο. Please go ahead, You can hear me, I assume, and I could hear you well. Λαγκάρτ. Εντάξει. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, κυρίες και κύριοι. Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι και πάλι εδώ ενώπιον της Επιτροπής σας για δεύτερη φορά σήμερα και δεύτερη φορά φέτος υπό την ε, αρμοδιότητά μου ως επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Τον Ιούλιο σας εξήγησα τις αρχικές επιπτώσεις της πανδημίας και σας εξέθεσα κάποιες δυσκολίες που υπάρχουν στο μην τραπεζικό τομέα. Τότε υπογράμμισα τις ε, αρμοδιότητε που έχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και σήμερα θα ήθελα να ξεκινήσω αναφερόμενοι στις δράσεις μας έκτοτε. Ήδη από τότε εξήγησε ότι ένα από τα προβλήματα τα οποία μας απασχολούσε ήταν το κύμα μείωσης της, πιστοληπτικής, της αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κλάδο. Έτσι λοιπόν, προχωρήσαμε σε μια ανάλυση ευαισθησιών για να δούμε ποια είναι η κατάσταση στην αγορά όσον αφορά ε, μεγάλες ποσότητες ε, ομολόγων τα οποία απολούνταν. Και εξετάσαμε διάφορα μοντέλα τα οποία συνδυάζουν μέτρα ποσοτικής ε, χαλάρωσης με επικάλυψη χαρτοφυλακίων, κάνοντας διάφορες υποθέσεις. Και φάνηκε ότι τέτοιες πωλήσει μπορεί να οδηγούν σε ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση, σε εντάσεις και είναι πρόβλημα και για την σταθερότητα. Η ανάλυση μας επίσης έδειξε ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα σε τομείς και σε χώρες. Όλα αυτά δείχνουν πόσο μεγάλη σημασία έχει η διατεωμιακή ε, αντιμετώπιση, όπως επίσης και μεταξύ χωρών κάτι το οποίο είναι και η κύρια αποστολή εξάλλου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, επίσης είπα ότι η μείωση των ε, τιμών ε, ενεργητικού συνοδεύεται και από μεγάλες πιέσεις για διάφορα funds και επιδεινώνεται έτσι η κατάσταση ρευστότητα στην αγορά. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου υιοθέτησε και σύσταση με την οποία ζητάει από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, την ΕΣΜΑ, να ασκήσει τις αρμοδιότητές της. Και με την κοινή αυτή δράση είπαμε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στα επενδυτικά funds, τα οποία επηρεάζονται κυρίως λόγω πανδημίας. Πρώτον, επενδυτικά funds που έχουν ανοίγματα σε εταιρικό χρέος και επίσης ε, τους παράγοντες εκείνους που δραστηριοποιούνται στην ε, αγορά στέγασης κατοικιών. Εντοπίσαμε λοιπόν διάφορες αδυναμίες οι οποίες θα πρέπει και να αντιμετωπιστούν. Πρώτον, κάποια funds έχουν κινδύνους ρευστότητας και αδυναμίες όσον αφορά τη διαχείριση της έλλειψης αυτής ε, ρευστότητας. Δεύτερον, μόνο λίγα funds έχουν διορθώσει τις διαδικασίες τους όσον αφορά την έλλειψη ρευστότητας. Η ΕΣΜΑ επίσης καθόρισε κάποια βήματα τα οποία θα πρέπει να αναλυθούν για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα έτσι ώστε τα funds να είναι καλύτερα προετοιμασμένα για μελλοντικά προβλήματα ρευστότητας και έτσι γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω την ΕΣΜΑ που αντέδρασε γρήγορα στις συστάσεις μας. Για το θέμα αυτό τώρα γενικότερα, τα επενδυτικά funds αποτελούν έναν όλο και πιο σημαντικό παράγοντα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον προηγούμενο μήνα δημοσίευσε την έκθεσή της σχετικά. Και πρέπει εδώ να σημειώσω ότι πολλοί από τους τομείς που εντοπίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου βρίσκονται έτσι κι αλλιώς στην διεθνή ατζέντα. Μεταξύ άλλων, πρόκειται για κινδύνους που έχουν να κάνουν ε, με την αγορά χρήματος και με τις ρομές ε, ροές που είχαμε στις αρχές της χρονιάς. Επίσης, ε, πήρε και κάποια μαθήματα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου από το Μάρτιο και τον Απρίλιο όσον αφορά τον τομέα των ασφαλίσεων. Έχω υπογραμμίσει σε επιστολή που έστειλα στον Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκι τα ζητήματα αυτά για να ενημερώσω για την αναθεώρηση της Solvency 2. Οπότε από την επιστολή αυτή δύο σημεία θέλω να αναφέρω. Πρώτον, κίνδυνη ρευστότητας. Σε αντίθεση με τις τράπεζες, το business model των ασφαλιστών δεν είναι το ίδιο. Δεν λαμβάνονται υπόψη κίνδυνοι με τον ίδιο τρόπο, η διαχειριστική κίνδυνοι μέσω παραγόγων που όμως μπορεί να αποτελέσουν πηγή εντάσεων όσον αφορά τη ρευστότητα. Όταν υπάρχει μεγάλη αστάθεια, όπως υπήρξε στις αρχές της χρονιάς, διαπιστώνουμε πολλές διαφορές όσον αφορά τις αποτιμήσεις. Κάτι το οποίο σχετίζεται βέβαια με ροές από τα ε, άλλα funds αγοράς χρήματος. Υπάρχουν επίσης μεγάλες διαφορές μεταξύ των αγορών. Γι' αυτό και πρέπει να ενισχυθούν οι απαιτήσει ρευστότητα στη Solvency 2 και οι επόπτες να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν κάποια διατήρηση προστασίας ρευστότητας και ένα συγκεκριμένο προφίλ ρευστότητας. Αυτό ήταν το πρώτο στην επιστολή. Το δεύτερο είναι ότι σε ορισμένες χώρες οι ασφαλιστές κατέληξαν σε ad hoc λύσεις για να βλύνουν τους τρισμούς και τις επιπτώσεις που είχαμε το Μάρτιο. Χρησιμοποίησαν λοιπόν μέτρα που είχαν στη διάθεσή τους, τα οποία όμως δεν είχαν σχεδιαστεί για αυτό το σκοπό. Τα μέτρα αυτά όμως δεν μπορούν να αντιστραφούν εύκολα και θα συνεχίσουν να προσφέρουν κεφαλαϊκή ανακούφιση για τα επόμενα δέκα χρόνια. Το αποτέλεσμα είναι η βελτίωση των αντικυκλικών μηχανισμών στην Solvency 2 και συμμετρικά μέτρα για ε, δημιουργία κεφαλαίου που να μπορεί να αντιδράσει σε περίπτωση απολειών σε δύσκολες αποχές. Τώρα, ποια είναι η εξολόγηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου όσον αφορά την αστάθεια και τα θέματα των τραπεζών. Η αναζωπήρωση του COVID-19, το δεύτερο κύμα δηλαδή, προφανώς και ενίσχυσε την αβεβαιότητα όσον αφορά την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ε, χρειάστηκαν λοιπόν μέτρα κατά τη διάρκεια της κρίσης, τα οποία στήριξαν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και επιτυχώς βοήθησαν να περιοριστεί να περιοριστούν οι επιπτώσεις της κρίσης. Όμως πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά τη ρευστότητά τους και χρεώνονται όλο και περισσότερο. Γι' αυτό όσο περισσότερο κρατήσει η κρίση, τόσο πιο δύναμη είναι και η ανάκαμψη και τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος ε, προβλημάτων στις τράπεζες και χροκοπίας. Αυτές οι αδυναμίες βέβαια παίρνουν χρόνο για να εντοπιστούν, για να εμφανιστούν και να επηρεάσουν τους ισολογισμούς. Το ίδιο ισχύει και για τις ε, συμφωνίες ε, αναβολής ε, πληρωμής χρέους. Γι' αυτό και χρειάζονται μέτρα, τα οποία σίγουρα όμως θα επηρεάσουν την κερδοφορία των τραπεζών. Η μετακύληση των κινδύνων στον δημόσιο τομέα οδηγούν σε μείωση της ποιότητας των κεφαλαίων που εμφανίζονται στους ισολογισμούς των τραπεζών. Τα δάνεια λοιπόν προς μη τραπεζικές ε, ε, μονάδες, όπως είπαμε και πριν, εμφανίζουν διαφορές από χώρα σε χώρα. Και ενώ ορισμένες κυβερνήσεις έχουν ήδη επεκτείνει την διάρκεια των εγγύσεων, παρόλα αυτά τα φαινόμενα κατακριμνισμού υπάρχουν ακόμα. Και ενώ οι τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο ανθεκτικέ μετά από την προηγούμενη οικονομική κρίση, οι προοπτικές όσον αφορά την ποιότητα του ενεργητικού υποβάλλεται σε πιέσεις για κερδοφορία και σε διαρθρωτικά προβλήματα, μεταξύ άλλων υψηλό κόστος και σε μερικές περιπτώσεις και σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τώρα το θέμα της ρευστότητας στις τράπεζες. 5% είχαμε το τελευταίο τρίμηνο του 19 και πήγε στο 2% στο δεύτερο τρίμηνο του 20. Και ενώ αυτό είχε να κάνει με τα δάνεια, παρόλα αυτά βρισκόμαστε σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που βρισκόμασταν σε προηγούμενες κρίσεις. Για να ξεπεράσουμε λοιπόν όσο γίνεται πιο ομαλά την κρίση, φυσικά και χρειαζόμαστε ένα υγιές τραπεζικό σύστημα. Και γι' αυτό είναι ζωτική σημασία για τις τράπεζες να αναγνωρίσουν και να φροντίσουν να προβλέψουν μέτρα σε περίπτωση που βρεθούν αντιμέτωπες με νέα κρίση. Πρέπει να δουν το θέμα των μη ξεπηρετούμενων ε, δανείων βέβαια, ε, αναδιάρθρωση δανείων, και άλλα μέτρα τα οποία θεωρούνται κατάλληλα. Η σημερινή κρίση μπορεί να αποτελέσει και μια ευκαιρία για να αντιμετωπιστούν κάποιε από τις μακροχρόνιες αδυναμίες του τραπεζικού τομέα, επιταχύνοντας την αναδιάρθρωση και την παγίωση. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό επίσης να χρησιμοποιήσουμε και διακράτηση των κερδών που συμπεριλαμβάνεται στα μέτρα πολιτική μα για να βοηθήσουμε την αντοχή των τραπεζών. Όπως θα θυμόσαστε, οι συστάσεις του Ιουνίου του 2020 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου μιλάει για κατανομή των ε, κερδών, ότι δεν πρέπει να δίνονται πόνους κλπ, τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο. Λαμβάνουμε υπόψη μας όλα τα επιχειρήματα υπέρ και κατά συνεχιζόμενης δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις σε όλους τους τομείς των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται σε συντονισμό με όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, άρα δηλαδή και με τη συμμετοχή των μακροπροληπτικών αρχών. Πριν ολοκληρώσω, θέλω να υπογραμμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου δεν έχει ξεχάσει τις μεσοπρόθεσμες προτεραιότητές του. Εντοπισμό δηλαδή των ατομικών φορέων και των συνδέσεων μεταξύ τους για να υπάρχει μια καλή χαρτογράφηση της κατάστασης, κάτι το οποίο είναι αναγκαίο για να μην υπάρχει μετάδοση των προβλημάτων παρετέρω. Χρειάζεται επίσης ομοιόμορφη αντιμετώπιση εκείνων των νομικών προσώπων που κάνουν τον εντοπισμό στην αγορά. Το τι μπορεί να κάνει ο μη ε, τραπεζικός τομέας είναι περιορισμένος. Χρειάζεται κάλυψη, κάποιοι τομείς αποκλείονται και πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα και γι' αυτό το ΕΣΚ έχει οθετήσει σύσταση όσον αφορά τον εντοπισμό των νομικών οντοτήτων. Έτσι, ζητάμε ένα νομικό πρέσιο το οποίο να εντοπίζει τις ε, νομικές αυτές οντότητες και τις συναλλαγές τους και να χρησιμοποιείτε το LEI πιο συστηματικά. Τελειώνω λέγοντας ότι τρέχουσα κατάσταση απαιτεί συνεχή στήριξη. Η ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση έδειξε πόσο σημαντική είναι η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ αυτών που αποφασίζουν την πολιτική σε όποιο επίπεδο και αν βρίσκονται. Πιστεύω ότι η δικιά σας συνεισφορά για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση ήταν ζωτική σημασία επίσης και ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις κοινέ μας προσπάθειε για να καταπολεμήσουμε την κρίση με ένα συνεχιζόμενο διάλογο. Αν το κάνουμε αυτό μαζί θα βρούμε τις κατάλληλες λύσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου μπαίνει στο δέκατο χρόνο λειτουργίας του και έτσι ετοιμάσαμε και την ένατη έκθεση δραστηριοτήτων μας. Θα συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε στην οικονομική σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει της εντολής μας. Ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω τώρα στη συζήτησή μας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε τον κύκλο απαντήσεων. Ήδη κανόνες, δύο λεπτά για ερώτηση, τρία λεπτά για την απάντηση. Η Ντανούτα Χούμπνερ από το ΕΛΚ ξεκινάει. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα, κυρία Λαγκάρτ. Μεγάλη χαρά που σας ακούμε. Ακούσαμε αυτά που είπατε. Όσον αφορά μακροπροληπτική δημοσιονομική σταθερότητα, τραπεζικός μη τραπεζικός τομέας, εξετάσατε προσεκτικά τα μαθήματα από το πρώτο κύμα του κορονοϊού και τι έγινε μέχρι τώρα. Ξέρω ότι υπάρχουν διαφορές και περιορισμένες αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ξέρετε τι βάρος έχει αβεβαιότητα στα όσα θα κάνουμε. Στο Ευρωκοινοβούλιο συζητούμε το πρόβλημα προσεκτικού εντοπισμού της σωστής απόσυσης των εκτάκτων υποστηρικτικών μέτρων για να αποφύγουμε αποτελέσματα που έχουν ε, πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Ποιους, πώς βλέπετε τους παράγοντες που θα καθορίζουν πότε πρέπει να αποσυρθούν τα έκτακτα ε, μέτρα από το σύστημα αυτό της ESRB και πώς μπορεί να υπάρχει σωστός αποτελεσματικός συντονισμός των διαφόρων διαδικασιών λαμβάνοντας υπόψη και διασυρωνιακές διαστάσεις στις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ χωρών αλλά και μεταξύ τομέων, όπως αναφέρατε. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χούμπνερ. Σωστά θέσατε τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Κρίσιμο σημείο απόφασης είναι αυτό για τις αρχές. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει σωστή διαχείριση του συστήματος, μπορεί να δημιουργηθούν κίνδυνοι σημαντικοί. Είπατε, σωστά. Απ' τη μια, έχουμε το αποτέλεσμα πολλαπλασιασμού. Cliff, όπως αναφέρατε. Και μετά, σε ανταπόκριση σε αυτό το κίνδυνο, πρέπει να τηρηθεί υποστήριξη ή να επεκταθεί, όπως είδαμε, σε κάποια σχήματα που εφαρμόζονται, κυρίως όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, τα μη ε, εξυπηρετούμενα δάνεια. Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε και έναν μελλοντικό κίνδυνο. Εάν διατηρηθούν επιμακρών τα μέτρα, τα έκτακτα, αυτό ε, δεν επιτρέπει τη σωστή διανομή του κεφαλαίου. και να διατηρηθούν μέσω των μορατόρια διάφοροι φορείς που από τη στιγμή που θα λήξει η πανδημία θα έπρεπε πιο αυτόνομα να διατηρούν την οικονομία. Είναι ένας κίνδυνος αυτός που αναφέρατε. Μην δημιουργήσουμε ένα τέρας. Επί, επί πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να διατηρούνται αυτά τα προγράμματα πλευράς δημοσιονομικής Γιατί η νομισματική πολιτική, τα ανέφερα αυτά στην προηγούμενη κουβέντα μας. Είπα ότι η σωστή νομισματική πολιτική, χαλαρή νομισματική πολιτική, στηριχτική θα πρέπει να διατηρηθεί όσο πλήττει η κρίση την οικονομία μας για να πετυχαίνουμε σταθερότητα τιμών. Τέλος. Ε, εστιαζόμεθα επί του αποφασιστικού σημείου αναστολής των μέτρων. Αυτό αφορά και το πώς θα γίνει η απόσυση της στήριξης. Ποιες είναι οι λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι σταδιακή εξάλληψη των μέτρων είναι καλύτερη προσέγγιση. Το είπα και η εισαγωγή. Χρειάζεται επίσης να δεχτούμε και να καλύψουμε τους κινδύνους από τα μη ε, εξυπηρετούμενα δάνεια που αντιμετωπίζουν, τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουν από τα κόκκινα δάνεια τράπεζες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενος, ο Άλφρεντ Σάντ από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ερώτηση. Η ερώτησή μου σχετίζεται με την ε, αξιολόγηση του ESRB τα χρόνια. Στην έκθεση του 2014 μέχρι το 2018 σε εκθέσεις, πάντα τονιζόταν 4-5 θέματα. όπως η, όπως η των αξιογράφων, αδυναμία των κλιματοστικών αγορών στον κόσμο. Η τελευταία αξιολόγηση του κινδύνου του Ιουνίου 2020 αντικατοπτρίζει τον αντίκτυπο του κορονοϊού. Αυξάνονται σε 7 οι κίνδυνοι. Ευρεία χρεοκοπία στον ιδιωτικό τομέα. Λόγω της ύφεσης, Πρώτο. Δεύτερο δύσκολη, δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον για τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείε και συνταξιωτικά συστήματα. Στο 2018 είπατε ότι αυτά είναι αποτελέσματα κυρίω από καιροποίηση αξιολογήσεως κινδύνων. Είναι κάτι παραπάνω από επικαιροποίηση. Εδώ βλέπουμε μεγάλη αλλαγή που ξεπερνά τα αποτελέσματα του COVID-19. Έχουμε και το θέμα του, το περιβαλλοντικό κλειδονισμών στην 7η θέση και προβλήματα στον κυβερνοχώρο. Αυτά δεν αφορούν το COVID-19. Τι έγινε και έχουν αλλάξει οι κίνδυνοι. Μειώθηκαν κάποιοι κίνδυνοι. Πώς δημιουργήθηκε η νέα ιεραρχία είναι το βασικό ερώτημα των κινδύνων. Ποια είναι η σχέση των νέων κινδύνων με αυτούς του παρελθόντος. Η αλλαγή έμφασης αντικατοπτρίζει μήπως κάτι άλλο. Η αλλαγή της ηγεσία στο συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο του ESRB περισσότερο από ότι η επιρροή της πανδημίας που άλλαξε λοιπόν η ιεράρχηση των κινδύνων. Κοιτάξτε με πρόεδρος του ESRB. Μπορώ να αναφερθώ μόνο στο πρόγραμμα του SRB. Προσεκτικότατα διαβάσατε, είναι σαφές αυτό και εντοπίσατε τους κινδύνους, τον κατάλογο κινδύνων της ένα της έκθεσης. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι οι παρόντες κίνδυνοι που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και θα αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον αυξήθηκαν από τους συγκεκριμένου που αναφέρατε και διαβάζω για να είμαι πιστή όπως και εσείς στο κείμενο, στην έκθεση. Έλλειψη, ρο, ε, μείωση, ε, ρίωση ε, ροή των κεφαλαίων και βάρο των χρεών που αυξάνεται, οπότε δεν μπορεί να συμμορφωθούν τα νοικοκυριά και επιχειρήσει στι ανάγκε. Αυτό προηγείται όλων των άλλων κινδύνων αυτή τη στιγμή. Να μην πούμε ότι άλλοι κίνδυνοι έχουν εξαλειφθεί και ότι δεν πρέπει να του προσέξουμε. Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να παρακολουθούνται και να του αντιμετωπίζουμε. Αλλά αυτό ο κίνδυνο συγκεκριμένο επικρατεί, κυριαρχεί. Δεύτερον, τα προβλήματα στο μη χρηματοστοτικό ιδιωτικό τομέα που δοκιμά την αντοχή των ευρωπαϊκών τραπεζών. Προσπάθησα να το εξηγήσω αυτό κάπως στην εισαγωγή μου, στα εισαγωγικά μου σχόλια, διότι είναι ένας κίνδυνος που πιθανότατα συλλογικά δεν είχαμε προβλέψει να παρουσιαστεί στο επίπεδο που παρουσιάστηκε, δηλαδή ότι η πίεση ήταν από τα επενδυτικά ταμεία ασφαλιστικές εταιρείε στις χρηματαγορές, κεντρικές τράπεζες τελικά, διότι έπρεπε να αντικαταστήσουμε εμείς και να προσθέσουμε ρευστότητα σε μια αγορά που κυρία βασικά είχε στεγνώσει. Αλλά υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι που αναφέρονται στην έκθεση, υφίστανται, θα συνεχίσει η ανάγκη να αντιμετωπίζονται και θα εξακολουθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Όσον αφορά το ESRB, σας διαβεβαιώνω ότι θα εξακολουθούμε να παρακολουθούμε την κατάσταση, να κάνουμε συστάσεις συναθρίζοντας όλους τους φορείς της αγοράς. Είτε για το θέμα εξυγίανσης, είτε για άλλα προβλήματα. Όλους τους τομείς της χρηματοπιστωτικής αγοράς θα τους συγκεράσουμε. Σας ευχαριστώ και τώρα το λόγο στον Λιγκαρικάνο από το Ρινιού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Λαγκάρτα. Σας ευχαριστώ για την προηγούμενη απαντήση σας. Το 2016 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν ένα από τα βασικά ε, στοιχεία για να έχουμε ε, μια σαφή μετάβαση σε μια ασφαλή κατάσταση. Αυτό έχει γίνει σχόλιο και από πλευρά μου και από το ESB και σε ό,τι αφορά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε μια πρόταση και μια ομάδα του Κοινοβουλίου πριν από κανένα χρόνο και τώρα με τις ιστορικές αυτές συμφωνίες για το 1-3 περίπου και για το Next Generation EU, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται λοιπόν στο, στη φάση που δημιουργεί μια εμβριονική φάση του ασφαλούς αυτού μέσου. Νομίζετε ότι η ESRB Ενδεχομένω να κάνει μια τέτοια συζήτηση και να αναθεωρήσει τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γαρικάνο για απάντηση. Και σημειώνω προφανώς τα δύο μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εισαγωγή δηλαδή ε, μιας ε, τυποποιημένης ε, ασφάλισης σε ό,τι αφορά τις σημεία έκθεσης που δεν εξυπηρετούνται και κατά δεύτερον να πούμε ότι σημειώνω ότι το Κοινοβούλιο θα ήθελε να δώσει τα χρήματα αυτά στο ESRB σε ό,τι αφορά συγκεκριμένη άμα ασφάλιση, αλλά να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου ήδη έχει τέτοια εντολή. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν με ένα dashboard κινδύνου για να δούμε τι είδου ανάλυση χρειάζεται για την συνεκτική και ασφαλή συλλογή δεδομένων προκειμένου θα να εκτιμήσουμε σωστά το τι θα γίνει στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά τώρα την ασφάλιση ε, μη εξυπηρετούμενων ε, ε, θέσεων, θέλουμε να μειώσουμε αυτές τις θέσεις και να έχουμε όμως ε, αρκετό κεφάλαιο, επαρκές κεφάλαιο σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα. Με ρωτάτε και δεν μπορώ να παραναπαντήσω ότι ναι, η Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κινδυνίου έχει κάνει προτάσεις στο παρελθόν και προφανώ ε, αυτέ οι προτάσει ε, καλωσορίζονται. Αλλά υπάρχουν πολύ σημαντικέ νέε εξελίξει. Και ένα ευρωπαϊκό ομόλογο. Το Next Generation EU ε προφανώς είναι ένα αποφασιστικό βήμα προς τη δημιουργία ευρωπαϊκών αποθεματικών, ασφαλών αποθεματικών Ξέρουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο απευθύνεται στην τρέχουσα κατάσταση, αλλά προφανώς και πλαισιώνει το, το πώς θα διαμορφώνονταν το ευρωπαϊκό safe asset. Και τέτοια στοιχεία πανευρωπαϊκής ε, ε, ε, κλίμακας είναι σαφές ότι τα θεωρεί ευπρόσδεκτα η αγορά. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο έχει η Λελένη Λαπόχτ από το ID. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λαγκάρτ, για την ακρόαση αυτή. Εγώ θέλω τη γνώμη σας για το ΤΕΦ, που εμπλέκουν συστημικούς κινδύνους, δεδομένου ότι πρόκειται για σύνθετα προϊόντα. και γίνονται ανταλλαγές σε αυτά. Τα σύνθετα τέτοια προϊόντα εγγυώνται μια περιορισμένη εγγύηση και μια απόδοση η οποία διασφαλίζεται από ένα swap, αλλά υπάρχει κάποια ελευθερία σε αυτόν που τα διαχειρίζεται και που δεν είναι ο εκδότης. Υπάρχει όμως ένας κίνδυνος εδώ αρκετά υψηλός, αν δεν προειδοποιηθεί ο τρίτος έγκαιρα. Το 98 είχαμε το LTSM που πτώχευσε και που οργάνωσε η Fed τότε τη διάσωση και μετά το 2011 πάλι που διάφοροι ρυθμιστές στράφηκαν ε, στα σύνθετα αυτά προϊόντα με ένα διπλό όμως κίνδυνο και για την εξασφάλιση και για το swap που μπορεί τελικά να μην απέδιδε. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν το εξή, κυρία Λαγκάρτ, πιστεύετε ότι αυτά το ΟΤΕΦ και κυρίως τα σύνθετα όντω μπορεί να είναι κίνδυνος εάν υπάρχει επένδυση από τρίτων που δεν συνδέεται άμεσα με, την, με το αρχικό προϊόν. Και έπειτα με τους δείκτες της αγοράς σε περίπτωση που υπάρχουν επενδύσεις σε τοπικά νομίσματα ή σε πρώτες ύλες. Δεν υπάρχει μεγάλη αστάθεια. Τέλος, η ρύθμιση η οποία επλαισιώνει τα σύνθετα αυτά προϊόντα καλύπτε, καλύπτει τις περιπτώσεις αυτές. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι το 2008 ήμουνα υπουργό Οικονομικών και μετά το 2011 ήμουνα επικεφαλής στο IMF, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μιλάτε για εξωτικές περιπτώσεις, προϊόντα κτλ. Όντως, κάθε φορά που ακούω τον όρο εξωτικά, είμαι επιφυλακτική. Εν πάση περιπτώσει. Εδώ πέρα πρόκειται για swaps, τα οποία φάνηκε να ήταν αρκετά ανθεκτικά στην αρχή της πανδημίας. Όμως, όταν υπάρχει επένδυση σε αγορές λιγότερο ρευστές, το Μάρτιο για παράδειγμα, είδαμε ότι έπεσαν τιμές στα EDF. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος που έχει εντοπιστεί και νωρίτερα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Πρόκειται για τον έλεγχο κινδύνου στο μη τραπεζικό τομέα, αλλά και από την Επιστημονική Επιτροπή που είναι αρμόδια για αυτά. Τώρα, σε τι βαθμό αυτή η αποσύνδεση είναι ανησυχητική και χρειάζεται παρετέρω εξέταση, οι μετοχές που συνεχίζουν να βρίσκονται σε διαπραγμάτευση ενώ αρχίζει κάποια ρευστοποίηση Μπορεί όμως να αντικατοπτρίζει και τους μηχανισμούς αρμπιτράζ. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το κατά πόσο TTF ε και τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία λειτουργούν και πώς μπορούν να δυσκολέψουν τη ζωή άλλων προϊόντων στις ε, χρηματοπιστωτικές αγορές. Σίγουρα θα πρέπει να το αποφύγουμε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και περνάμε στον επόμενο. Για Κελίνας, από τους Πρασίνους, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Λαγκάρτ, να σας συγχαρώ για την δέσμευσή σας αυτούς τους δύσκολους καιρούς και στη σημερινή συζήτηση. Δεν είναι απλά όλα αυτά για σας. Να αναφερθώ στα αρνητικά επιτόκια. Τα οποία μπορεί να παραμείνουν ε, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν και σε άλλες ακροάσεις και στην προηγούμενη ακροάση. αλλά βλέπετε να υπάρχει κάποιος αντίκτυπος στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, στις τράπεζες, στα ταμεία συνταξιευότητας κτλ. Σε ό,τι αφορά τα επιτόκια. Και δεύτερο τμήμα της ερώτησης, τι γίνεται σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Θα υπάρξουν θεσμικές επιδράσεις γιατί είναι εύκολος ο δανεισμός, πιο εύκολος ο δανεισμός ε, σε σχέση με την ε, μεταρρύθμιση. Αλλά αυτό ενδεχομένω να οξύνει το πρόβλημα. Και τη μεταφορά του κινδύνου στον καταναλωτή ενδεχομένω σε ό,τι αφορά τα συνταξιωτικά προϊόντα. Και αυτό αποτελεί μια πηγή ανησυχίας. Το κόστος επίσης ε, θα μπορούσατε παρακαλώ να σχολιάσετε σε ό,τι αφορά δηλαδή τις άμεσες επιδράσεις των επιτοκίων και οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις του περιβάλλοντος αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήταν λίγο εισαγωγικά. Να πω ότι από πλευράς της ΕΚΤ και ζητώ συγγνώμη που δεν απαντώ ω ε, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου το κάνω αυτό, αλλά από πλευρά τη ΕΚΤ σαφώ υπάρχει σαφή εμπειρία σε ό,τι αφορά τα αρνητικά επιτόκια. Ξέρω εγώ ότι ακούγεται λίγο περίεργο. Νομίζω ότι ο τρόπο που ε, χρησιμοποίησαμε τα αρνητικά επιτόκια για να πετύχουμε το στόχο μα ήταν αποτελεσματικό. Επίση, το σύστημα κατηγοροποίησης το οποίο δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο πέρσι, επίσης ε, αποδέχτηκε να είναι αποτελεσματικό για να εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν ε, υπερβολικά αποθέματα σε επίπεδο τραπεζών και ότι θα υπήρχε κάποια προστασία σε αυτό το επίπεδο. Αλλά τώρα να βάλω το καπέλο μου ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου προφανώς και Διαρκώς αναλύουμε τον αντίκτυπο των χαμηλών επιτοκίων σε όλους τους τομείς του οικονομικού συστήματος, όχι μόνο στο τραπεζικό σύστημα. Και η κίνδυνη για την δημοσιονομική σταθερότητα σε ό,τι αφορά τα αρνητικά αυτά επιτόκια, θεωρούμε ότι μπορούν να κατηγοροποιηθούν σε τρεις κατηγορίες. Καταρχάς, η χαμηλή απόδοση που θα επηρεάσει την ε, ανθεκτικότητα των φορέων. Κατά δεύτερον, η ε, κίνδυνη που παίρνουν τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και τρία των ε, διευθυντικές αλλαγές στο σύστημα. Κοιτώντα λοιπόν τους διάφορους τομείς, οι ασφαλιστικές, τα μία συνταξιοδότηση, τα αναφέρατε και τα δύο, έχουν προβλήματα να τα βγάλουν πέρα. Φερεγγιότητας, τα μοντέλα λοιπόν, ε, τα επιχειρησιακά των ε, εταιρεών αυτών είναι πολύ ευάλωτα σε χαμηλά επιτόκια και επίσης έχουμε και τον συνολικό αντίκτυπο των χαμηλών ε, επιτοκίων σε ό,τι αφορά την κερδοφορία των τραπεζών. Αυτό ακόμα συζητιέται γιατί υπάρχουν και παράγοντες ε, αντιστάθμιση όπως η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το ανέφερα αυτό και προηγουμένως. Και βλέπουμε λοιπόν ε, στοιχεία ανάληψης μεγάλων κινδύνων από χρηματοπιστωτικά εντρέματα για να προσφέρουν συστήματα συνεισφορών και να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο προς τους καταναλωτές. Μας δείχνουν λοιπόν οι αναλύσεις μας αύξηση των εκθέσεων σε εναλλακτικές ε, κατηγορίες κινδύνων Άρα εκτιμούμε τους κινδύνους αυτούς και τους παρακολουθούμε στενά. Και αυτό και σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται στην παρούσα φάση, μεταξύ άλλων και στον τομέα των ασφαλιστικών με το Solvency 2. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή. Eugene Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο, Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω το εξή. Η εμπειρική γνώση λέει ότι όταν επιμένουν τα αρνητικά επιτόκια δημιουργούν στεγαστικές φούσκες. Μία από τις μελέτες δείχνει την σχέση αυτή που φάνηκε στις χώρες όσα το Βέλγιο, Φιλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και άλλες χώρες τα τελευταία έξι χρόνια όλες αυτές οι χώρες της Ευρωζώνης κατέγραψαν μεγάλες αυξήσεις στα επιτόκια υποθηκών. Στη δικιά μου χώρα, στην Σλοβακία, η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική των πρόσφατων ετών οδήγησε σε φαινόμενο που θα μπορούσε να ονομαστεί η Σλοβακική Στεγαστική Επανάσταση δημιουργείται στρέβλωση στην αγορά με αύξηση των τιμών στέγασης. Δεν υπάρχουν κατοικίες διαθέσιμες και αναγκάζονται οι αρχές να παρέμβουν με ρυθμίσεις, με περιορισμούς ε, στα ενίκια κλπ. Κύριε Λαγκάρτ, η δικιά μου ανησυχία είναι οι παρενέργειες της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ που μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη παρέμβαση των δημοσίων αρχών τελικά. Η κυρία Λαγκάρντα, ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας που έχει να κάνει με το στεγαστικό κλάδο. Ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου ε, παρακολουθεί στενά αυτό το ζήτημα. Το 2017 και το 2019 δημοσιεύσαμε μελέτες για αυτόν τον κίνδυνο, το στεγαστικό, και κάποιες προειδοποίησεις μάλιστα και συστάσεις για διάφορες χώρες. Και δημοσιεύσαμε επίσης και έκθεση για τις αδυναμίες που υπάρχουν σε άλλους μεσητικούς κλάδους πέρα της στέγασης. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό και για τους Ευρωπαίους οι οποίοι είναι ιδιοκτήτε μια κατοικία, αλλά και γενικότερα για την οικονομία. Συνεπώ, το 2021, κατά πάσα πιθανότητα, θα υπάρξει νέα μελέτη για τη στεγαστική κατάσταση, αλλά προς το παρόν οι τιμές φαίνεται να έχουν αντισταθεί στις επιπτώσεις της πανδημίας χάρη στα στηρικτικά μέτρα τα οποία έχουν υιοθετηθεί με διάφορα προγράμματα και όπως είπατε και εσείς και χάρη στα χαμηλά επιτόκια. Οπότε, ο κύκλος αυτός, κατά τη γνώμη μας, θα επιβραδυνθεί κάπως. Κυρίως οι αρνητικές μακροοικονομικές επιπτώσεις. Και θα οδηγηθούμε σε μεγαλύτερη απασχόληση. Οπότε, αυτές οι κυκλικές ε, δραστηριότητες και επιπτώσεις επηρεάζονται φυσικά από αδυναμίες διερθρωτικές κάτι το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα η στέγαση να γίνεται πιο δύσκολη. Όλα αυτά έχουν υπογραμμιστεί και έχουν να κάνουν με τη χρηματοπιστωτική κατάσταση, αλλά έχουν να κάνουν και με την προσφορά. Και σε μερικές χώρες η προσφορά είναι πολύ περιορισμένη. Γιατί είτε δεν υπήρχαν προγράμματα κοινωνικής κατοικίας ή γιατί είναι πολύ περιορισμένα και έτσι θα έλεγα ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου πάντα πρόσεχε τους κινδύνους στο στεγαστικό κλάδο και θα συνεχίσουμε. Και σίγουρα είναι κάτι το οποίο αφορά όλους τους Ευρωπαίους. Ευχαριστώ πολύ. σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πρέπει να πω στους συναδέρφους ότι σταματάει η διερμηνία γιατί τελείωσε ο χρόνος μας. Παρόλο που έχουμε κάποιους ομιλητές ακόμα, δίνω το λόγο στο Γιώργιο Κίρτσο, πρώτα απ' όλα από το ΕΛΚ. Mr. Kyrtsos, please go ahead. Press the speak button. Chair, maybe we go to the next speaker and we come back yes. to Mr. Kyrtsos.